Voilà, nous allons commencer notre session de lapres λοιπόν, έχουμε το σημείο 17 της ημερήσιας διάταξης. Ε, είναι σημαντικό επίσης σημείο. Αποτελεί το θέμα μας αυτό το προτινόμενο παναφρικανικό πρόγραμμα στα πλαίσια του μέσου αναπτυξιακής συνεργασίας και της κοινή στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αφρικής. Ξεκινήσαμε αυτή τη συζήτηση χθε το απόγευμα, είναι το Παναφρικανικό Πρόγραμμα, το οποίο προτείνει η Επιτροπή και αυτό μέσω μιας, ε, ε, ενός καινούριου μέσου αυτής της συνεργασίας. Και έχουμε μια περιληπτικό κείμενο σχετικά με αυτό το πρόγραμμα και για τη σχέση με την κοινή στρατηγική Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αφρικής. Έχουμε από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Διαχείρισης Αναπτυξιακής Πολιτικής τον κύριο Σερίφ, τον εκπρόσωπο και η κυρία Τισή κανονικά. Ο κύριος, ο κύριος, συγγνώμη, ο κύριος Τισή. Δεν είναι κύρια, είναι κύριος ο Τισή. Οι οποίοι θα μας πούν ε, ποιες είναι οι συστάσεις τους μετά από τις αναλύσεις τους. Επίσης τον κύριο Ίγκε, το εύχομαι το καλό ορίσατε που είναι ο επικεφαλής της μόνιμης αντιπροσωπείας ε, της, ε, από την Αφρικανική Ένωση στην ε, Ευρώπη, στις Βρυξέλλες. Και τον ευχαριστώ. Σημαντικό δεν είναι για μας να ακούσουμε και τις απόψεις των Αφρικανών εταίρων μας πάνω στο σχέδιο αυτό. Και αυτό πριν να ξεκινήσει η όλη διαδικασία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Προσπαθούμε να ψηλαφίσουμε την κατάσταση, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Έχει μεγάλη σημασία αυτή η κοινοβουλευτική διάσταση αυτή τη κοινή στρατηγική στην οποία και προωθούμε. Τον κύριο Γκάλερ επίσης ε, καλέσαμε, ο πρόεδρος της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που έχει να κάνει με τις σχέσεις με το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο. Τον ε, καλέσαμε να συμμετάσχει στη συζήτηση, δεν είναι ακόμα εδώ, δεν παρίσταται, αλλά έχουμε, τρέφουμε ελπίδες ότι θα μας έρθει σε λίγο. Οι εμπειρογνώμονες μας λοιπόν έχουν το λόγο από 10 λεπτά ο καθένας. Βέβαια διαλέξτε εσείς ποιος θα λάβει πρώτος το λόγο. Ευχαριστούμε. Um, thank you very much uh, for this invitation. Ευχαριστώ πολύ για την ε, πρόσκληση να απευθυνθώ στην Επιτροπή Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα σας δώσω λίγες πληροφορίες υποβάθρου για ορισμένα από τα κύρια ε, στοιχεία που αναφέρονται και στο έγγραφο που σας έχουμε μοιράσει για το Παναφρικανικό Πρόγραμμα και την κοινή στρατηγική Αφρικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα προσπαθήσω να εστιαστώ στα κύρια σημεία του και κυρίως στον τρόπο με τον οποίο ε, σχετίζεται με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τη συζήτηση για το μέσο αναπτυξιακής συνεργασίας. Πρώτα απ' όλα, ε, λίγα στοιχεία για το κέντρο μας. Το Κέντρο Διαχείρισης Αναπτυξιακής Πολιτικής. Να σας παρουσιάσουμε τι είμαστε. Το Παναφρικανικό Πρόγραμμα Καμιά φορά αναφέρεται στα αγγλικά ω ΠΑΠ που είναι ατυχέ αυτό γιατί ε, το ίδιο ακρονίμιο χρησιμοποιείται για το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο. Το κέντρο μα λοιπόν, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Διαχείριση τη Αναπτυξιακή Πολιτική, ε, έχει ένα ε, μνημόνιο συνεργασίας με την Αφρικανική Ένωση. Έχουμε εκπροσώπους χωρών της Αφρικής και της Καραϊβικής. Και από το 2007 και ακόμα και πιο πριν εξετάζουμε τα ζητήματα που αφορούν στις ε, σχέσεις, ε, εταιρικές σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αφρικής. Γι' αυτό λοιπόν θεωρήσαμε σημαντικό να σας ε, αποστείλουμε αυτό το έγγραφο ανάλυσης του προτινόμενου Παναφρικανικού προγράμματος. Το πρώτο ζήτημα. Γιατί χρειάζεται ένα Παναφρικανικό πρόγραμμα. Θεωρώ ότι ένα από τα σημαντικότερα ε, ζητήματα που ε, βρίσκουμε είναι ότι δεν υπάρχουν ικανοποιητικοί χρηματοδοτικοί μηχανισμοί για την στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ Αφρικής και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό έχει ε, θεωρηθεί το αγκάφι στις σχέσεις μεταξύ των δύο υπηρών. Και θεωρούμε ότι δύο, η Αφρική και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αξιοποιήσουμε τον καλύτερο τρόπο αυτή την εταιρική του σχέση. Αυτό επίσης αποτελεί ε, και στοιχείο που βλάπτει την ε, αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο συγκεκριμένο θέμα. Η στρατηγική σχέση θεωρούμε ότι δεν τίθεται ένα αμφιβόλο η θεμελιώδης αξία της ωστόσο έχει δώσει μέχρι στιγμής μικρή προστιθέμενη αξία. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν και να εξευρεθούν οι πόροι οι οποίοι ε, θα δώσουν ε, την ουσία, την, στην πράξη της εταιρική αυτής σχέσης. Και το Παναφρικανικό πρόγραμμα μπορεί να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Μία από τις κριτικές που ακούγεται για την κοινή στρατηγική είναι ότι δεν έχουν υπάρξει ε, απτά αποτελέσματα, ε, υλοποιηθήσεις ενέργειες. Και η ίδια στρατηγική και το πρόγραμμα μάλλον έχει τα δικά του ε, θέματα, προβλήματα, αλλά θεωρούμε ότι θα οδηγήσει σε απτά αποτελέσματα, ιδίω στον τομέα της ειρήνης και της ασφάλειας. το Παναφρικανικό πρόγραμμα επίσης θα βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει την Αφρική ως μία ενιαία ήπειρο, κάτι το οποίο παλαιότερα υπήρξε πρόβλημα κατά την υλοποίηση της κοινή στρατηγικής Αφρικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πού βρισκόμαστε λοιπόν σήμερα. Υπάρχει μια ε, ε, πρόταση για ένα δισεκατομμύριο ευρώ σε χρηματοδοτικό μηχανισμό για προγράμματα περιφερειακά και σε επίπεδο υπήρου ε, το, το οποίο είναι, ε, είναι χρήματα τα οποία μπορούν να ενταχθούν στον ΤΑΚ. Η ανταπόκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφέρεται, ε, λέει μάλλον ότι το 90% αυτών των κονδυλίων θα μπορούσαν να ενταχθούν στον ΤΑΚ. Υπάρχει, ΤΑΚ υπάρχει λοιπόν μια μικρή διαφορά εδώ. Αλλά η συνένεση του Παναφρικανικού Κοινοβουλίου η υφίσταται ήδη. Είναι η συγκεκριμένη χρονική στιγμή πολύ σημαντική γιατί η επόμενη σύνοδος μεταξύ ε, Αφρικής και Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ε, φτάσει μέχρι το 2000, θα, δεν θα γίνει παρά μόνο μετά το 2014. Έτσι λοιπόν η επόμενη σύνοδος κορυφής θα μπορέσει να θα, μπορούσε να ξεκαθαρίσει ορισμένα στοιχεία της στρατηγικής, της κοινής στρατηγικής και μετά από αυτή να προκύψει και η χρηματοδότηση. Αλλά ένα ζήτημα είναι ότι θα πρέπει να καταλήξουμε στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο πιο πριν, επομένως πρέπει να σκεφτούμε με ποιον τρόπο μπορούν να διασφαλιστούν τα κονδύλια του Παναφρικανικού Προγράμματος στο πολιτες δημοσιονομικό πλαίσιο. Ποιε είναι λοιπόν οι ευκαιρίε και οι κίνδυνοι που έχουμε μπροστά μας. Θα βοηθήσει, ε, χωρί αμφιβολία, τις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωση και Αφρικής και σε διπυρωτικό και σε ε, επίπεδο ε, υπήρου. Το πρόβλημα της έλλειψης πόρων πάντα ήταν σημαντικό και προκειμένου να είναι αξιόπιστη η κοινή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προκειμένου να υπάρξουν και αυτά τα αποτελέσματα χρειάζονται ε, αυτοί οι πόροι, οι κίνδυνοι. Τους αναφέρουμε πάρα πολύ ξεκάθαρα στο έγγραφό μας ε, και αυτοί οι κίνδυνοι ε, ξεφεύγουν από το ζήτημα των χρημάτων. Η στρατηγική σχέση ε, έχει προβλήματα τα οποία ξεφεύγουν από το ζήτημα των κονδυλίων. Το ε, Παναφρικανικό πρόγραμμα μπορεί να συνεισφέρει, αλλά δεν μπορεί φυσικά να λύσει όλα αυτά τα ε, προβλήματα. Μπορεί να υποστηρίξει, μπορεί να δημιουργήσει μια ορμή, έτσι ώστε να, να συμβούν. Σε περίπτωση που δεν υλοποιηθεί όμω το Παναφρικανικό πρόγραμμα, πιστεύω ότι άνθρωποι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στην Αφρική θα αρχίσουν να αμφισβητούν κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διατεθειμένη να ε, χρησιμοποιήσει, να αποδώσει τους ε, πόρους που χρειάζονται για τη στρατηγική τη σχέση με την Ήπειρο. Εάν οι πόροι που διατίθενται είναι περιορισμένοι, ίσως δοθεί εντύπωση ότι δεν λαμβάνουμε με σοβαρότητα το θέμα. Τα... Οι πόροι από το μέσο της αναπτυξιακής συνεργασίας ε, μπορούν να αξιοποιηθούν και αυτό φαίνεται και στην πρόταση της Επιτροπής αλλά και στην, στο προσχέδιο ε, της απάντησης του Κοινοβουλίου. Λοιπόν, μπορεί με, χρησιμοποιώντας το Παναφρικανικό πρόγραμμα να υπάρξει διάλογος μεταξύ των δύο υπήρων, η μία υπήρος και η άλλη ε, ενωμένε. αλλά θα μπορέσει επίση να δώσει και τη δυνατότητα η συζήτηση να περάσει πέρα από τα ζητήματα αναπτυξιακή συνεργασία. Τίθεται επίση το ζήτημα πώ θα συνεχιστεί το πρόγραμμα μετά από το 2020. Υπάρχει το ε, θέμα του κατά πόσον θα ενταχθεί στον προπολογισμό. Ο αντίκτυπο αυτού του προγράμματο λοιπόν στις σχέσεις της Αφρικής με την Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω την ανέφερα, θα αυξήσει την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κοινή στρατηγική ε, εξάλλου όταν είχε δημιουργηθεί η αντίληψη μας ήταν ότι θα ήταν κοινή η ευθύνη για την χρηματοδότηση των προγραμμάτων. Δηλαδή ότι θα είναι ισότιμη εταίρη η Αφρική και Ευρωπαϊκή Ένωση στα προγράμματα που εντάσσονται σε αυτή τη στρατηγική. Πιστεύουμε λοιπόν ότι το Παναφρικανικό πρόγραμμα μπορεί χωρίς να λύνει τα θεμελιώδη ζητήματα να προσδώσει ε, μια μεγαλύτερη δυναμική στη στρατηγική σχέση. Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου λοιπόν τώρα και της ε, ε, κοινή αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου στο, στην Αφρικανική έχει σχέση κυρίως με τον δημοκρατικό έλεγχο. Πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει δημοκρατικός έλεγχος αυτή τη στρατηγική σχέση; Πρώτον υπάρχει η δυνατότητα να ενταχθούν αυτές οι δράσεις στο πλαίσιο της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας του Συμβουλίου. Επίσης το Κοινοβούλιο μπορεί να ε, εξασφαλίσει ότι θα υπάρχει συνοχή με άλλα χρηματοδοτικά μέσα, καθώς επίσης και να λειτουργήσει το Κοινοβούλιο ως θεματοφύλακας ευρωπαϊκών αξιών. Εμείς θεωρούμε από την πλευρά μας ότι προκειμένου το πρόγραμμα να είναι ε, κοινό, θα πρέπει να υπάρχει σεβασμός στον διάλογο με τους εταίρους από την Αφρικανική Ήπειρο. Και με τον ίδιο τρόπο που το πρόγραμμα μπορεί να συνεισφέρει στην ειρήνη και την ασφάλεια στην Αφρική, με τον ίδιο τρόπο θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε το πρόγραμμα για να υποστηρίξουμε ε, πρωτοβουλίες ε, στις οποίες η Αφρικανική Ένωση έχει αναπτύξει πρότυπα, για παράδειγμα στα ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου. Υπάρχει λοιπόν ένα διάλογο που πρέπει να λάβει χώρα μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Αφρικανική Ένωση στο ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τώρα συμπερασματικά. Η κοινή στρατηγική αποτελεί ένα ε, καλό πλαίσιο, αλλά πρέπει να δοθεί μια νέα δυναμική σε αυτό και αν δεν το κάνουμε τώρα πότε θα το κάνουμε. Ε, τα μέσα είναι απαραίτητα, δεν είναι όμως, δεν αρκούν από μόνα τους. Μπορούμε να δώσουμε περισσότερους σπόρους, αλλά ε, όπως ε, λένε, εάν ε, έχουμε ένα αυτοκίνητο που δεν δουλεύει καλά, ακόμα και να του βάλουμε περισσότερη βενζίνη δεν θα αρχίσει να τρέχει πιο γρήγορα. Λοιπόν, αλλά απ' την άλλη, ακόμα και αν δεν δίνουμε πόρους, δεν πρόκειται να υπάρξει βελτίωση. Άρα η κατάσταση έχει ως εξή. Έχουμε ένα πλαίσιο το οποίο πρέπει να βελτιωθεί. Το Παναφρικανικό πρόγραμμα θα βοηθήσει σε αυτήν την βελτίωση. σε όλα τα θεσμικά όργανα και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να εργαστούν προ την κατεύθυνση τη βελτίωση τη στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ ε, Αφρική και Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η χρηματοδότηση πρέπει να λειτουργεί συμπληρωματικά προς την πολιτική ε, καθοδήγηση και τον πολιτικό διάλογο έτσι ώστε να καταλήγουμε σε από κοινού προτεραιότητες. Και πάλι τίθεται το ερώτημα πώς μπορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συνεργαστεί με το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο έτσι ώστε να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και αν υπάρχουν ερωτήσεις με χαρά θα τις απαντήσω ε, και στα πιο επιμέρους ζητήματα στα οποία δεν είχα το χρόνο να μπω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μήπως θα θέλατε κάτι να συμπληρώσετε κύριε Τησί. Μερικά σχόλια να προσθέσω ε, για να συμπληρώσω την εξαιρετική κατά τα άλλα παρουσίαση του συναδέλφου. Το πρώτο, η κοινή ε, φύση της εταιρική σχέσης. Θα πρέπει και οι Αφρικανοί να δεσμεύσουν περισσότερα κονδύλια σε αυτή την εταιρική στέση Και σήμερα υπάρχει ένα διέξοδο και δεν βοηθάει από την αφρικανική πλευρά. Ελπίζω να λυθεί το συντομότερο. Κάτι άλλο που μπορεί να σας φανεί ευκαταφρόνητο η ε, λεπτομέρεια, το είπε και ο Άντριος στην αρχή. Δεν υπάρχει περαιτέρω ε, χώρος για να αλλάξει το ΠΑΠ, να το πούμε ΠΑΦ επειδή είναι παναφρικανικό πρόγραμμα και το, το, ΠΑΠ, το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο λέγεται ήδη ΠΑΠ. Δεν μπορεί το πρόγραμμα να έχει το ίδιο όνομα. Δεν ξέρω, ίσως αυτό να σας φανεί, είπαμε, δευτερεύον, αλλά είναι ένα ζήτημα. Αυτά από πλευρά μου και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ακούσουμε τον κύριο Χίγκε που θα μας ε, δώσει ενδεχομένως την άποψη της Αφρικανικής Ένωσης για το θέμα αυτό και να απαντήσει στο πολύ εύστοχο ερώτημα. Εάν βάλουμε περισσότερη βενζίνη σε ένα σαράβαλο θα λειτουργήσει καλύτερα. Merci, Madame la ναι, κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ. Χαίρομαι ιδιαίτερα που πέρα το λόγο για να ανταλλάξω μερικά πράγματα σχετικά με αυτήν την μεικτή πολιτική, κοινή πολιτική Ευρωπαϊκή Ένωση και Αφρική και για θέματα τη χρηματοδότηση του σχεδίου δράση στρατηγική. Αυτή η εταιρική σχέση μεταξύ των δύο είναι ειδική φύσεως και γι' αυτό για αρκετές πτυχές οι σχέσεις μεταξύ των δύο επίρων χρονολογούνται από πάρα πολύ παλιά και αυτό έχει διαμορφωθεί από την ιστορία, τη γεωγραφία και καταφυλίγει σε μορφές συνεργασίες και στην πολιτική και στην οικονομική, στρατιωτική, κοινωνική, πολιτιστική και γλωσσική επίσης από το 2000 στη διάσκεψη του Καΐρου ε, ξεκίνησε μια πολιτική ώστε να συνδυαστούν, συγχωνευτούν όλα αυτά με μια κατάλληλη συνεργασία στα πλαίσια μιας κοινή στρατηγικής που να βασίζεται σε ένα διάλογο ανάμεσα στις δύο υπήρους που να είναι υπέρ και των δύο και θα είναι μια σημαντική πρόοδος αυτή υιοθέτηση μια κοινή στρατηγική στη Λισαβόνα το 2007 ε, το Σεπτέμβριο δείχνει μια νέα εποχή στις σχέσεις μεταξύ των δύο υπήρων. Αυτή η εταιρική σχέση βασίζεται σε μια κοινή ενόρεση και των δύο δηλαδή, κάτι το ενισχυμένο και μια εμβάθυση επίσης της συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα που βασίζεται πληρωμικά σε, πάνω σε βασικές αρχές και σε σαφείς στόχους. Αυτό το νέο πλαίσιο συνεργασίας προσφέρει ταυτόχρονα και αρκετές δυνατότητες, αλλά δημιουργεί και πολλές προκλήσεις. Όσον αφορά τις δυνατότητες, η συνεταιρική αυτή σχέση μεταξύ των δύο αποτελεί μια πραγματική δυνατότητα για κάθε ήπειρο ξεχωριστά σε, κάθε, σε ένα κόσμο που είναι αλληλεξαρτώμενος. Και με τους δύο έχουμε ακριβώς 82 χώρες που συμμετέχουν και πρόκειται για ένα σημαντικό στοιχείο της παγκόσμιας γεωπολιτικής και στα Διεθνή Φόρουμ και με την οθέτηση κοινών θέσεων σε σημεία κλειδιά κοινού ενδιαφέροντος και επίσης για θέματα που έχουν να κάνουν με το μέλλον του πλανήτη οι προκλήσεις ε, πώς τίθενται σε μας ε, σχετικά με τις ελπίδες που γεννιούνται από αυτή την κοινή πολιτική και έτσι να οδηγήσουμε, να μεταφράσουμε σε συγκεκριμένες πράξεις αυτή την όρεση και να έχουμε κατάλληλες ενέργειες στην εταιρική αυτή σχέση. Τώρα για την εφαρμογή του πρώτου σχεδίου δράσης ε, με κύρια προσοχή στι κύριες προκλήσεις, αλλά τα πράγματα κάπως αρνητικά σχετικά με το ρυθμό εφαρμογής ε, και μπορούμε να πούμε σαν παράδειγμα ότι δεν προσυπέγραψαν ακριβώς, ε, μάλλον δεν συμφώνησαν με την αρχή αυτή να είναι μία ενότητα η Αφρική και με τη συνεργασία όλων αυτών των δύο. Η συνεργασία καθορίζεται από μεμονωμένες συμφωνίες, κάτι που δεν είναι υπέρ της συνοχής. Για να πετύχουμε όμως αυτό, καταλαβαίνουμε ότι απαιτείται χρόνος και σιγά σιγά θα το πετύχουμε. Επίσης, ανάμεσα στις προκλήσεις είναι ότι δεν υπάρχουν σχέσεις ανάμεσα στις επαφές μεταξύ των πυρογνώμων και σε τοπικό, σε περιφερειακό επίπεδο. Δεν υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στην πολιτική διάσταση και στην ε, πτυχή ανάπτυξης της εταιρική σχέσης και ότι χρειάζεται ακόμα περισσότερο να συμμετάσχουν όλοι εκείνοι οι αρμόδιοι σε αυτή την κοινή στρατηγική, κυρίως το Κοινοβούλιο, η Περιφερειακή Οικονομική Επιτροπή, η ε, φορείς ε, από διάφορες πλευρές ε, και επίσης ε, για τα χρήματα που απαιτούνται για το πρόγραμμα δράσης στα πλαίσια της κοινή αυτής στρατηγικής. Πέντε χρόνια μετά από την υιοθέτηση αυτής της στρατηγικής, τι γίνεται σήμερα. Πρέπει να ενισχυθεί το όραμα των εταίρων γιατί όλα αυτά εξαρτώνται από τη δυνατότητα να πετύχουμε αποτελέσματα, απτά αποτελέσματα και όπως σας είπα να γίνει κάτι το συγκεκριμένο, ο κάθε στόχος, εντάξει φιλόδοξος εταιρική σχέσης που να ανταποκριθεί στις προσδοκίες αυτού του νέου πλαισίου συνεργασίας. Τώρα τι θέλουμε να εξετάσουμε σήμερα. Είναι η πτυχή η παναφρικανική. Γιατί αυτή η πτυχή παναφρικανική, επαναλαμβάνω. Τα κονδύλια που έχουμε ε, μεταξύ του πρώτου και δεύτερου προγράμματος δράσης κυρίως προέρχονται από το δεύτερο ΦΕΝΤ ακριβώς και θα δείτε ότι ε, όταν δόθηκαν τα χρήματα κονδύλια από το δεύτερο ΦΕΔ το 2006, η κοινή στρατηγική ακόμα συζητιόταν και το Σεπτέμβριο του 2007 υιοθετήθηκε στη Λισαβόνα και ε, μια πτυχή ακριβώς παναφρικανική ε, προωθείται αυτό από μακρύ χρονικό διάστημα, σιγά σιγά υιοθετείται και μετά από τη δήλωση της Λισαβόνας το 2007 και μετά είχαμε και πάλι μια διάθεση που επιδείχθηκε για να συμμετάσχει ο καθένας στην κοινή στρατηγική και όλα αυτά εμφανίζονται στις σημαίες διατάξεις των συναντήσεων μεταξύ των δύο μερών σε κάθε επίπεδο. Για ένα οικονομικό μέσο τώρα για την κοινή στρατηγική ε, πρώτα καθοδηγούμεθα από τα εξή κίνητρα. Σύμφωνα με το ότι θα πρέπει να ευθυγραμμιστούμε για μια αποτελεσματική βοήθεια όπως ζητείτε και όπως διατυπώνεται εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα και έτσι η αφρικανική πλευρά θα μπορούσε να συμμετάσχει πλήρως στον όλο προγραμματισμό των δραστηριοτήτων για τις οποίες ε, θα εξυπηρετήσουν ακριβώς τα χρήματα αυτά. Και αυτή η κοινή στρατηγική θα, θα πρικοδοτηθεί και με τα κατάλληλα κονδύλια για ένα καλό προγραμματισμό, σωστό προγραμματισμό και για να εξασφαλιστεί η μακροβιότητα αυτής της στρατηγικής. Και ακόμα επίσης πρόκειται αυτή η κοινή στρατηγική να πρικοδοτηθεί με κατάλληλα κονδύλια για την ε, σχετική πολιτική και θεωρώ ότι τα χρήματα και το αφρικανικό πρόγραμμα θα έχει να κάνει με τη, σχέση 2000, με τη, με τη περίοδο 2014-2020 που θα καλύψει ε, το, από το 2014 μέχρι το 2016 και από το 2017 μέχρι το 2019 καθώς και το 20, δηλαδή δυόμιση περίπου προγράμματα δράσης. Καταλαβαίνετε ότι είναι σημαντική αυτή η χρηματοδότηση για το όλο σύνολο από τις οκτώ εξωτερικές σχέσεις της κοινή στρατηγικής ε, εκείνο που πάει καλύτερα είναι αυτό που έχει να κάνει με την ασφάλεια και αυτό πώς εξηγείται κύριος ότι υπάρχουν κατάλληλα απαραίτητα κονδύλια όπως προγρέπονται στο δεύτερο φέντε στο σε πέντε και σας το είπα αυτό δείχνει καθαρά ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με κονδύλια ανεπαρκή. Και εδώ πάντα κύριε Πρόεδρε σε αυτό που ρωτήθηκε πριν από λίγο, δηλαδή ότι ε, όλοι μας θα είμαστε υπεύθυνοι ή για την επιτυχία ή για την αποτυχία αυτής της κοινή στρατηγικής. Έχουν περάσει μόλις πέντε χρόνια από τα νιώθια η στρατηγική αυτή, εντάξει είναι και λίγο και πολύ εκείνο που λένε και υπάρχουν άλλοι που λένε ότι έγιναν πολλά, άλλοι που λένε λίγο και ακριβώ για μια αρχιτεκτονική ε, θεσμική νομίζουμε ότι πάνω σε αυτό υπάρχουν πράγματα που μπορούν να βελτιωθούν και η πρόκληση σημερινή τι θα γίνει με την τρίτη διάσκεψη του χρόνου, πώς ακριβώς θα προσθέσουμε μπροστά στους ε, ηγέτες κρατών και κυβερνήσεων και για το 2020 τι θα έχουμε υλοποιήσει γιατί πρέπει να δούμε τα συγκεκριμένα που έχουν γίνει και να είναι κάτι το απτό αυτή η εταιρική σχέση εμφανίζονται αρκετέ δυσκολίε, όχι εμπόδια, όλα δυσκολίε τέλο πάντων, και θα μπορούμε να ξεπεράσουμε μαζί μέσα ενό κοινού διαλόγου, αλλά η χρηματοδότηση αποτελεί σημαντικότατη πτυχή, αποτελεί σημαντικό κρίκο τη αλυσίδα για να προχωρήσουμε σε αυτή τη συνεργασία και πρόκειται για μια σημαντική πρόκληση για να προχωρήσουμε, γιατί χωρί καύσιμο δεν μπορούμε ούτε καν να διορθώσουμε το όχημά μα. Τι να την κάνουμε τη βενζίνη, αν δεν πηγαίνει ο κινητήρα. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω λόγο στον κύριο Μπέρμαν, που είναι συγητή μα για το συγκεκριμένο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ως συγητή σα για το DCI, το Μέσο αναπτυξιακή συνεργασία, πρέπει να σας πω ότι εξεπλάγει λίγο όταν είδα αυτό το μικρό εδάφιο για το Παναφρικανικό πρόγραμμα ένα δισεκατομμύριο και οι δράσεις που ορίζονται χωρούσαν σε μια σελίδα και λιγότερο. Ωραίο αυτό το παιχνιδάκι σκέφτηκα για να παίξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χωρίς να έχει και πολλούς περιορισμούς, δράσεις ε, συγκεκριμένα περιγεγραμμένες. Έχω λοιπόν τις αμφιβολίες μου. Και χρειάστηκε λίγο να το μελετήσω μετά γιατί μου μπήκαν ψήλοι στα αυτιά. Βεβαίως συμφωνούμε όλοι και υποστηρίζουμε την ιδέα ενός ξεχωριστού χρηματοδοτικού μέσου για να ε, υλοποιήσουμε την ατζέντα μας με την Αφρική και είναι σημαντικό και χρειάζεται βεβαίως να έχει την απαραίτητη πρικοδότηση για να λειτουργήσει καλά. Και επανειλημμένα το Κοινοβούλιο ζητούσε ένα τέτοιο χρηματοδοτικό μηχανισμό σε προηγουμένα του ψηφίσματα. Αλλά Όπως ε, είπαν ε, οι εμπειρογνώμονες και ο εκπρόσωπος της Αφρικανικής Ένωσης, υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι που συνδέονται εδώ με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν μου επιτρέπετε να κάνω κάποια σχόλια. Το DCI, ο ΜΑΣ δηλαδή, Μηχανισμός για την Αναπτική Συνεργασία, είναι ένα εργαλείο ανάπτυξης και η Επιτροπή μας εδώ πάντα επέμενε σε αυτό τον ειδικό στόχο. Είναι ειδικού σκοπού ο μηχανισμός. Η μείωση και κρίζωση της φτώχειας. Η στόχη της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας. Σε αυτή την παράδοση εγγράφεται και η δική μου να προβλέπεται η ένταξη στον ΤΑΚΤ, στην Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας αλλά εδώ η στρατηγική αυτή βάζει τα θεμέλια για μια εταιρική σχέση που υπερβαίνει κατά πολύ βεβαίω την αναπτυξιακή συνεργασία και την εκρίζωση της φτώχειας. Εγώ δεν το αμφισβητώ αυτό, το αντίθετο μάλιστα. Αλλά έχουμε επίσης την ευθύνη να προστατεύσουμε ε, την ίδια τη φύση του μηχανισμού αναπτυξιακής συνεργασίας. Θα πρέπει να βρούμε στο μέλλον παραπληρωματικούς, συμπληρωματικούς, όπως είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, το μέσο εταιρική σχέσης, για τομείς ε, συνεργασίας που εκφεύγουν της αναπτυξιακής και δεν έχουν σχέση με την μείωση και κρίζωση της φτώχειας. Δεύτερον, για την κοινή στρατηγική μας με την Αφρική είναι και παραμένει μια κοινή προσπάθεια που να βασίζεται στην αρχή της πλήρους και ισότιμης θέσης. Το DCI, το ΜΑΣ, είναι ο μηχανισμός αυτός μονομερής. Ε, τον ορίζουν οι Ευρωπαίοι νομοθέτες, τον ορίζουν το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο και τον προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο εσωτερικός μας κανονισμός και οι κανόνες δεν μας ε, επιτρέπει να ε, αντιγράψουμε ε, όσα έχει τη συμφωνία του Κοτονού. Είναι άλλη ιστορία της ΑΚΕΕΦΤΗ. Και το Παναφρικανικό πρόγραμμα έχει προτεραιότητες χρηματοδότησης που από κοινού ορίζονται με τους Αφρικανούς εταίρους και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να έχουμε ε, αυτή την ε, πολυτομεακή προσέγγιση και να συμμετέχουν οι πάντες. Τα κοινοβούλια και το Παναφρικανικό, το είπατε κι εσείς, και άλλοι ενεχόμενοι. Οι δικές μου τροπολογίες έχουν ακριβώς αυτό το στόχο. Και παραθέτω από το άρθρο 13α της νέα τροπολογία μας, θα πρέπει να βασίζεται στο διάλογο και να ε, ειδωθεί στο πλαίσιο της κοινή στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, να συμμετέχουν όλοι οι ενεχόμενοι συμπεριλαμβανομένου του Παναφρικανικού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, στο τέλος των ε, διαπραγματεύσεων λοιπόν. Και ποιοι θα πρέπει να είναι βασικά οι τομείς συνεργασίας. Αυτό είναι το δυσκολότερο. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αφορά την κοινή στρατηγική Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αφρικής με πρόγραμμα δράσης, χωρίς να μπαίνει και σε πολλές λεπτομέρειες. Αλλά τα προγράμματα δράσης που τρέχουν τώρα λήγουν το 2013. Ενώ το μέτρο αναπτυξιακή συνεργασία είναι μέχρι το 2020 και το PAP επίση. Και η επόμενη σύνοδος κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικής θα λάβει χώρα του χρόνου και μπορεί να επανεξισορροπήσει τις προτεραιότητες. Θα ήταν καλό να έχουμε καλύτερη περιγραφή λοιπόν των τομέων συνεργασίας στο παράρτημα 6 ε, του DCI, του, ε, του ΜΑΣ. Θα κάνω και άλλες τροπολογίες σε αυτές τις γραμμές για το μέσο αναπτυξιακή συνεργασία, αλλά θα πρέπει να έχουμε αρκετή ευελιξία για να ε, ανταποκρινόμαστε σε αλλαγή προσανατολισμών που θα έχουμε συμφωνήσει πολιτικά από κοινού. Δηλαδή, Χρειάζεται αφενός νομοθετική σαφήνεια αφενός και από την άλλη ε, ε, σεβασμός για την αρχή ε, του ownership, αυτό που λένε τη ιδιοκτησία του εγχειρήματο. Θα πρέπει να φτάσουμε σε αυτή τη σαφήνεια και σε αυτή την ειλικρίνεια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, η Πρόεδρος. Ο κύριος Γκέρενς έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εδώ ε, ίσως ε, απομακρυνθεί πάρα πολύ αυτή η συζήτηση με αυτόν τον τρόπο, γιατί η τάση είναι να δείχνομαι και αυτοί που απ' έξω παρακολουθούν τη συζήτησή μας δεν θα καταλάβουν τίποτα. Πάρα πολλές εταιρικέ σχέσεις, συνεχώς περισσότερες ε, και αυτές οι εταιρικέ σχέσεις ανταποκρίνονται σε μία ανάγκη είναι πρωτοπόρες ε, για μια προστιθέμενη αξία. Η μεγάλη προστι... σημαντική προστιθέμενη αξία σε αυτή την εταιρική σχέση είναι πώς ε, θα απέναντι από τον ορισμό τον αρμόδιο που είναι μια τίγρης χάρτινη ε, που προωθούσε τους δικτάτορες των αφρικανικών χωρών εδώ βαθίζεται σε κάτι το θεωρητικό που ευτυχώς ε, αναφέρεται και εξηγείται ε, χάρτα της Αφρικανικής Ένωσης για την ασφάλεια στην Αφρική ε, είναι κάτι το ιδιαίτερο πρωτοποριακό, δηλαδή ότι δεν είναι κανείς αδιάφορος, όχι να μην αναμειχθεί, αλλά να μην διαφερθεί και έτσι ορισμένοι αναπτύσσονται όπω όπως πρέπει στα πλαίσια αυτής της τουρκικής σχέσης με μια μεσολάβηση όπου δεν μπορούμε να τους κερδίσουμε και οι αγγλόφωνοι Αφρικανοί καταφέρουν να έχουν αυτή τη διαμεσολάβηση ε, και σε γαλλόφωνες ε, σχέσεις ε, χώρες ακόμα όπως την ακτή ελεφαντεστού και έτσι και να οργανώσουν ένα μέρο ασφαλείας τους και μάλιστα ιδιαίτερα αποτελεσματικά και στην αρχή του δεκαετία του 2000 ε, το συζητήσαμε αυτό για να δούμε εάν θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε στη χρηματοδότηση ενός μέρους της οργάνωσης της ασφάλειας ε, στην Ήπειρο αυτή μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης. Και είχαμε πει τότε ότι ήταν ε, προσωρινή μένα αλλά καλή καλή πρωτοβουλία, κάτι που θα έπρεπε να έχει και πολιτικό χαρακτήρα απ' έξω και νομίζω ότι εκτός από τη χρηματοδότηση ε, όλα αυτά ανταποκρίνονται σε μια πραγματική ανάγκη. Τι με ανησυχεί κάπως τώρα εμένα είναι αυτά τα εισαγωγικά που ακούσαμε και που τόνισαν τους κινδύνους μέσω πολλών εταιρικών σχέσεων. Τώρα δεν καλό καταλαβαίνουμε ποιος κάνει τι η ιταλική σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αφρικής ε, με χρηματοδότηση από το DCI γεωγραφικά ε, για τα κράτη είναι οι χώρες ΑΚΕ μείον ε, χώρες Καραϊβικής, μείον του Ειρηνικού, αλλά μαζί με τις Βόρειας Αφρικής. Είναι λοιπόν μια ενότητα που αδιαχώριστη, εντάξει, καλό αυτό, αλλά μπερδεύονται τα πράγματα όταν αυτά αποτελούν πια μια πραγματικότητα από τα γεγονότα για τους ιδιαίτερους άξονες τους πολιτικούς. Τι έγινε σε περιφερειακό επίπεδο η ασφάλεια, εκεί είναι το πρόβλημα. Εκεί είναι ότι δεν μπορεί να προχωρήσει αυτό σε περιφερειακό επίπεδο γιατί η Επιτροπή φαίνεται πια καθαρά η τάση της ότι προωθεί αυτές τις εταιρικές σχέσεις και αυτό συζητήθηκε με την Αφρικανική Ένωση και κυρίως με, με αυτούς που συμμετέχουν σε περιφερειακό επίπεδο η Οικονομική Επιτροπή των ε, Κρατών της Ανατολικής Αφρικής, ε, όπου βλέπουμε ότι με την οργάνωση εμπορίου ακριβώς δεν πάνε καλά τα πράγματα. Εταιρικέ οικονομικές σχέσει δεν προχωράνε αυτές και για την οργάνωση της ασφάλειας. τα απ' όλα δεν υπάρχουν ε, ε, κονδύλια και δεν νομίζουμε ότι μέσα στην DCI θα μπορέσει να υπάρξει αποτελεσματική χρηματοδότηση. Ποιο είναι ο κίνδυνος επίσης να περιμένουμε, περιμένουμε προσδοκίες πολλές και να μην υπάρξει μια συνέχεια. Με δοθεί μια συνέχεια μετά θα πρέπει να δούμε ακριβώς για το διάλογο αυτό, ε, να δούμε για τον ΕΠΑΤ. Εδώ ήταν εργοτάξιο θεσμικό στην Αφρική αλλά υπάρχουν ορισμένα κενά, κάτι μαύρες τρύπες. Εδώ η Ευρώπη κινδυνεύει να χάσει το δρόμο της αυτές τις εταιρικές σχέσεις. Ακούσα μια φράση, τι είπατε. Η εταιρική σχέση στον τομέα αυτό, εάν αποτύχει, δεν ξέρω, αυτό κατάλαβα εγώ. Δεν θα είχε δυνατότητα η Ευρώπη να βαρύνει στην όλη πολιτική, άσκηση πολιτικής μεταξύ των δύο υπήρων. Αλλά έχουμε το γύρο οργανισμό που είναι οι χώρες ΑΚΕ και 20 άλλες εταιρικές σχέσεις μεταξύ των κρατών μελών. Και αυτό προώθησαμε το πολύ καλό δηλαδή ε, μάλλον αυτό το που, δεν είναι, που είναι αρνητικό, ότι αν πετύχουμε στον τομέα θα πετύχουμε παντού. Όχι, τι γίνεται με τους υπόλοιπους. Νομίζω ότι τα πράγματα θα πρέπει να παρουσιάζονται περισσότερο συγκεντρωμένα ακριβώ για τις προσπάθειες που καταβάλουμε, που δεν είναι μόνο η στρατηγική μας μέσω αυτής της εταιρικής σχέσης, αλλά και μέσω εταιρικών σχέσεων ε, μέσω της των ΑΚΕ και μια τελευταία παρατήρηση για τις χώρες ΑΚΕ. Και εκεί αναρωτιέται κανείς για το μέλλον ε, με τις ε, σχέσεις με τις χώρες ΑΚΕ. Ναι, πρόκειται για απτό κίνδυνο και με απασχολεί με αυτό το θέμα ε, και το ερώτημα τι θα γίνει με το μέλλον των, των χωρών ΑΚΕ. Έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο, μια φάση σκέψης που δεν αποκλείεται πια και η εξαφάνιση αυτής της, της σχέσης με τις χώρες ΑΚΕ. Και θα ήταν ε, αρνητικό αυτό. Και ακούσαμε και το πρόβλημα για το πώς εντάζεται στον προπολογισμό του ΦΕΔ και είπατε τι θα γίνει, σε ποιο σημείο ακριβώς βρισκόμαστε τώρα και είναι απλή απάντηση. Δεν ξέρω αν δεν προχωρήσουμε περισσότερο από τα τελευταία 40 χρόνια, τα τελευταία, τότε δεν κάνουμε τίποτα. Αυτό έστω και για αυτό τον ενταχθεί στον προπολογισμό μέχρι το 2020, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Τότε θα έχουμε και νέες προτάσεις και τι θα ήθελα να σας πω. Σημαντικά είναι όλα αυτά αλλά μην ξαναδημιουργήσουμε από την αρχή τον όλο μηχανισμό, την όλη αρχιτεκτονική της εταιρικής, των εταιρικών σχέσεων μεταξύ Ευρώπης και Αφρικανικής Ένωσης. Α, και για το πού βρισκόμαστε ερώτημα και αυτό. Αυτό ε, με αυτές τις υποθέσεις, με αυτή τη θετική σχέση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και αναφερθήκαμε στους νέους που συμμετέχουν στα πλαίσια της Συμφωνίας του Κοτονού από την κοινωνία των πολιτών, ιδιώτες με νέα εταιρική σχέση, αλλά δεν ακούμε και πολλά να λέγονται για αυτό το European African Business Forum. Και μετά στην ε, περίοδο Καντάφη δεν ακούσαμε πια να γίνεται λόγος για αυτά. Ευχαριστώ. Δίνω το λόγο στον εαυτό μου. Για να πω το εξή. Αυτό που με ανησυχεί σε αυτό το μέσο, το DCI, το Μηχανισμό Αναπτυξιακής Συνεργασίας, είναι η πλευρά που ονομάζεται εταιρική σχέση, η πλευρά που ονομάζεται διάλογος, αλλά και πολιτικός διάλογος μεταξύ των κοινοβουλίων. Μα γνωρίζουμε τι δυσκολίε έχουμε για να ε, αναγνωριστεί ο λόγος του Κοινοβουλίου στο DCI, ότι θα έχουμε λόγο Κοινοβούλιο στα στρατηγικά κείμενα. Εκεί να δείτε τι συζήτηση έχει να γίνει και πόσο έντονες οι συζητήσεις θα είναι τους ερχόμενους μήνες. Και πρέπει να σας πω ότι και στην εταιρική σχέση με την Αφρική, αν χρησιμοποιήσουμε αυτό το μέσο, θα έχουμε αυτές τις δυσκολίες. Και με κάνει να φοβούμε ότι θα είναι ένα μέσο στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περισσότερο παρά στη διάθεση των κοινοβουλίων. Και θα ήθελα εδώ να με διαφωτίσετε, αν μπορείτε, από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Euh, θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Euh, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτέ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον κύριο Χίγκερ για την παρέμβασή του και του κύριο Περλάν, καθώς και όλους τους άλλους ευρωβουλευτές και το κέντρο του ECDPM που μας έκανε αυτή την παρουσίαση που κατά έναν τρόπο ε, αποτελεί συνέχεια μιας εξέλιξης της ανάλυσης των αποτελεσμάτων αυτής της εταιρικής σχέσης. Στην αρχή ε, λειτουργήσαν ως, ε, διευκόλυναν την συζήτηση την... και στη συνέχεια παρακολούθησαν την εξέλιξη της υλοποίησης αυτής της εταιρικής σχέσης και με χαρά βλέπω ότι τώρα το ECTPM καλείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να παρουσιάσει το πλαίσιο μέσα στο οποίο διεξάγεται ο διάλογος για το Παναφρικανικό μέσο. Ε, το ερώτημα του κατά πόσο είναι δικαιολογημένο αυτό το μέσο επειδή το αυτοκίνητο μας έχει βλάβει σχετίζεται με την εξή εικόνα που θα ήθελα να σας δώσω. Έχουμε δύο αυτοκίνητα. Το ένα είναι αυτό που προσπαθούμε από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ε, επισκευάσουμε και έχει σχέση με την χρηματοδότηση και η άλλη, το άλλο αυτοκίνητο έχει σχέση με την αφρικανική πλευρά και με την ασφάλεια. Το Παναφρικανικό πρόγραμμα, του οποίου το όνομα μπορούμε να αλλάξουμε αν είναι απαραίτητο, ε, θεωρώ ότι εντάσσεται σε ένα πολύ συγκεκριμένο ιδιαίτερο πολιτικό πλαίσιο, το οποίο ε, ήδη είχαμε ε, προβλέψει ε, και δημιουργήσει το 2007 στη Λισαβόνα. Είναι μια πολιτική προσέγγιση από τη μία ήπειρο στην άλλη. Είναι μια προσέγγιση βάσει της οποίας εμείς βλέπουμε την Αφρική ως μία ενιαία ήπειρο και θεωρώ ότι θα είναι χρήσιμο ένα εργαλείο το οποίο θα λειτουργήσει ως το κέντρο βάρους όλων των πρωτοβουλειών που αναπτύσσονται μεταξύ των δύο υπήρων. Και γιατί αυτό, γιατί αυτή η στρατηγική εταιρική σχέση είναι μία από τις επτά στρατηγικές σχέσεις που αναπτύσσει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τον υπόλοιπο κόσμο και είναι η μόνη στρατηγική σχέση που απευθύνεται ε, σε μία ήπειρο και η οποία δεν έχει ένα συγκεκριμένο ε, ειδικό χρηματοδοτικό μέσο. Η Επιτροπή θεωρεί λοιπόν ότι είναι, ε, έχει έρθει η ώρα να, να βάλουμε μαζί όλα τα, τα, τα σχετικά κονδύλια και όλες τις σχετικές χρηματοδοτήσεις, ακόμα και αν το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν ανταποκρίνεται σε όλα τα προβλήματα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η σύνοδος κορυφής ε, που θα γίνει στο τέλος του 2013 αρχή 2014 μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αφρικής θα πρέπει να είναι ένα φόρουμ στο οποίο όλοι οι συμμετέχοντες θα εξηγήσουν, θα δείξουν κατά πόσον είμαστε διατεθειμένοι να συνεχίσουμε αυτή την εταιρική σχέση έτσι ώστε το 2015 να φτάσουμε ε, σε ε, έναν κόσμο με 2,7 δισεκατομμύρια ε, ανθρώπους οι οποίοι θα πρέπει να συνεπάρξουν. Έχουμε όλες αυτές τις εξελίξεις στην ε, Αφρική. Έχουμε την Αραβική Άνοιξη. Και παρόλα αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει στη διάθεσή της ένα χρηματοδοτικό μέσο ή μια συγκεκριμένη στρατηγική ώστε να ανταποκριθεί στις κοινέ προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ένωση και η Ήπειρος της Αφρικής. Ξέρω ότι με κύριε Μπέρμαν, θα ήθελα να σας δώσω ορισμένα παραδείγματα τομέων στους οποίους το παναφρικανικό ε, πρόγραμμα θα είχε προστιθέμενη αξία σε σχέση με αυτό που ήδη έχουμε. Όλοι αναφερθήκατε σε, άλλα, ε, ε, σε άλλους μηχανισμούς, του Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, στον Μηχανισμό Γειτονίας, άλλους μηχανισμούς του προπολογισμού. Αλλά όσον αφορά την εταιρική σχέση, το Παναφρικανικό πρόγραμμα θα μας έδινε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε ζητήματα που έχουν χαρακτήρα διεπιρωτικό. Θα μπορούσαμε... Αντιλαμβάνομαι μάλλον τις επιφυλάξεις που εξέφρασε ο κ. Μπέγμαν σε σχέση με τον ΜΑΣ, αλλά η εταιρική σχέση μεταξύ Αφρικής και Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, είναι μια σχέση κοινού ενδιαφέροντος που πηγαίνει πέρα από την ανάπτυξη. Αλλά ε, για να σας δώσω λοιπόν αυτά τα παραδείγματα, τα συγκεκριμένα, τι θα μπορούσε να δώσει περισσότερο ένα παναφρικανικό πρόγραμμα. Θα σας αναφέρω τρία παραδείγματα. Το πρώτο, σε σχέση με τον διάλογο και τη συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, Αφρικανικής Ένωσης στο ζήτημα της διακυβέρνησης, της ασφάλειας και της ανάπτυξης. Θεωρώ ότι έχουμε ένα προκαθορισμένο πλαίσιο το οποίο μας επιτρέπει να εργαστούμε αποτελεσματικά και όχι αφηρημένα. Είναι ένα νέο πλαίσιο το οποίο γνωρίζουμε και το οποίο δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να αξιοποιήσουμε από κοινού. Είναι η αφρικανική αρχιτεκτονική διακυβέρνηση. Είναι μια αρχιτεκτονική διακυβέρνηση η οποία μοιάζει λίγο με αυτό που κάνουμε στον τομέα της ειρήνης και της ασφάλειας, που αποτέλεσε αντικείμενο διαλόγου μεταξύ ημών μέχρι στιγμή και δημιουργήθηκε και μια σχετική πλατφόρμα. Ένα συγκεκριμένο λοιπόν παράδειγμα. Η Αφρική υιοθέτησε μια χάρτα για τη δημοκρατική διακυβέρνηση και τις εκλογές. Αυτό οδηγεί σε δράσεις οι οποίες δεν θα μπορούσαν να υλοποιηθούν σε εθνικό ε, ή ε, απλώς περιφερειακό επίπεδο, αλλά χρειάζονται ε, συζήτηση και διάλογο σε επίπεδο υπήρου. Να λοιπόν που θα μπορούσε να βοηθήσει ένα παναφρικανικό πρόγραμμα. Δεύτερον, η συνέχιση της συνεισφορά μας στην αρχιτεκτονική για την ειρήνη και την ασφάλεια Έχουμε καλύψει πολύ ε, δρόμο και έχουμε καταφέρει να βρούμε την σύνδεση μεταξύ ασφάλειας και ανάπτυξης. Τα υπάρχοντα μέσα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης θα μπορούν να συμπληρωθούν με δράσεις διαλόγου επί του θέματος της ασφάλειας και της ειρήνης είτε σε διεπηρετικό επίπεδο ή σε επίπεδο υπήρου. Και το τρίτο παράδειγμα, η κινητικότητα και η απασχόληση, η οποία ταιριάζει απόλυτα με τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, ιδίω ε, με το πρόγραμμα για την αλλαγή, για την, τη νέα στρατηγική για την ανάπτυξη στον τομέα της οικονομικής ανάπτυξης, στον τομέα της ε, απασχόλησης. Και εδώ μπορούμε να έχουμε μια προστιθέμενη ε, αξία ε, εάν υπάρξει συνεργασία σε επίπεδο υπήρων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αφρικανικής Ένωσης. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, να δοθούν κίνητρα σε μικρές επιχειρήσεις, έτσι ώστε να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας Υπάρχει επίσης το ΚΑΝΤΕΠ, ένα ε, πλαίσιο το οποίο είναι γνωστό στο αφρικανικό διάλογο ε, και είναι ένας διάλογος στον οποίο συμμετέχει ο τομέας της γεωργίας, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό. Και τέλος, στο επίπεδο της ενοποίησης περιφερειακής ε, σε επίπεδο υπήρου ή ε, Ίσως είναι υπερβολικά ισιόδοξο ο στόχος του να το καταφέρουμε μέχρι το 2017 είναι να δημιουργηθεί μια ε, ζώνη ελεύθερων ανταλλαγών που θα πηγαίνει πέρα από τις διαπραγματεύσεις για τις εταιρικές σχέσεις και που θα εξυπηρετήσει τα κοινά συμφέροντα Αφρικής και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει επίσης το ε, πρόγραμμα ε, για τις υποδομές, ε, για την ανάπτυξη υποδομών στην Αφρική, που θα μπορούσε να βοηθηθεί. Έτσι λοιπόν, η συνεργασία για τα κοινά μας συμφέροντα αυτών των δύο εταίρων ε, θα, φαίνεται ακόμα, θα γίνει ακόμα περισσότερο ερατή όταν αναφερόμαστε σε ζητήματα που είναι παγκόσμιες προκλήσεις, όπως για παράδειγμα η τρομοκρατία, η αλλαγή του κλίματος, το περιβάλλον. Θα σταματήσω εδώ λοιπόν την αναφορά μου σε συγκεκριμένα παραδείγματα. Αλλά κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ε, προσθέσω και σε αυτό που ανέφερε ο κύριος Μπέρμαν, χρειάζεται να υπάρξει ε, μια εργασία πάνω στην πρόταση. Το ζήτημα της κυριότητας, το ζήτημα του κατά πόσον ε, από κοινού θα διαχειριζόμαστε το, το πρόγραμμα. Ε, όπως και σε ένα μουσικό σύνολο, κανείς δεν μπορεί όπως γενικά στο πλαίσιο της ε, κοινή ε, Στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωση Αφρικής κανείς δεν μπορεί να ε, δουλέψει μόνος του. Πρέπει να δουλέψουμε από κοινού. Χάρη λοιπόν σε αυτό το μηχανισμό, στο πλαίσιο των αρχών στις οποίες όλες συμφωνήσαμε στην Τρίπολη και στη Λισαβόνα, για μια εταιρική σχέση που επικεντρώνεται στους πολίτες, στους δημοκρατικούς θεσμούς. Το γεγονό ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο αναπτύσσουν όλο και πιο ε, στενές ε, σχέσεις, θεωρώ ε, πως θα πρέπει να το ενισχύσουμε και ο Παναφρικανικός Μηχανισμός θα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Κλείνοντας, άκουσα κάποιες επιφυλάξεις σε σχέση με τη διαδικασία του Κοτονού αφενός και αφεντέρου τη δημιουργία νέων μηχανισμών. Δεν, θεωρώ ότι και οι δύο πρωτοβουλίες είναι συμβατές μεταξύ τους. Δεν, δεν βλέπω γιατί να υπάρχει σύγκρουση το 2020 πιθανώς θα χρειαστεί να αναθεωρήσουμε κατά πόσον είναι ε, συμβατή η εταιρική σχέση όπως θα έχει εξελιχθεί με την ε, Σύμφωνη του Κοτονού. Αλλά αυτό το παναφρικανικό πρόγραμμα θα μπορούσε να λειτουργήσει ως καταλήτης για την εξέλιξη της σχέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρική σε κάθε περίπτωση αυτό το χρηματοδοτικό μέσο δεν θα είναι το, η μόνη λύση για να λύσουμε όλα τα προβλήματα της εταιρική μας σχέσης. Φυσικά θα χρειαστούν και πολιτικές λύσεις. Αλλά η, μια πολιτική στρατηγική εταιρική σχέση πρέπει να ανταπο... αντανακλάται και σε ένα τέτοιο μέσο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που να συνεχίσουμε το τη συνάντησή μας. Ε, θα ήθελα να χαιρετήσω Ευρωπαίους πολίτες από τον Ράιδαρ Θα ήθελα να τους ε, ευχηθώ μια ημέρα ενδιαφέρουσα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τη Ρινανία Παλατινάτο, η προσκεκλημάνη μας εδώ, μιλάμε για τη σύσταση ενός νέου μέσου παρέμβασης, το καταλαβαίνετε, για το σύνολο της Αφρικανικής Υπήρου. Σας ευχόμαστε λοιπόν ε, ε, καλή επικοδομητική μέρα σε όλους. Τώρα ο συνάδελφος Μπέρμαν που αποτελεί από τους τηλοβάτες εδώ της Επιτροπής μας, ο οποίος και θα απαντήσει σε αυτά που μας είπε η Επιτροπή. Κύριε Πρόεδρε, αυτός ο στήλος, ο πυλώνας θα κατεδαφιζόταν εάν δεν μπορούσαν όλοι αυτοί εδώ οι πολίτες οι Ευρωπαίοι με την υπέροχή τους βοήθεια, στήριξη που στηρίζουν το ευρωπαϊκό σχέδιο και που μας βοηθούν να προχωρήσουμε για κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο τώρα εδώ αυτή την εποχή αλλά παντού όλα αυτά αποτελούν τη βάση του ευρωπαϊκού σχεδίου οι πυλώνες πραγματικά. Τους ευχαριστούμε λοιπόν που έρχονται. Είναι πολύ καλή αυτή πρωτοβουλία που σας προσκάλεσαν που ήρθατε από τη Ρωανία Παλατινάτο. Να πω κάτι τώρα για το πολιτικό πλαίσιο αυτό. Φαίνεται καθαρά ότι είναι συμφέροντος ευρωπαϊκού η Αφρική να μπορεί να είναι ικανή να λύσει τα δικά της τα προβλήματα. Ισχυρή πολιτική Ευρώπη και μια Αφρικανική Ένωση που να μπορεί να δράσει. Και Πώς, πώς το λέμε στα γαλλικά. Στα γαλλικά πώς το λέτε, πώς το λέτε αυτό το Pan-African Program, αυτό το παναφρικανικό πρόγραμμα ακριβώ, αν μπορεί να στραφεί προς αυτήν την κατεύθυνση και να ενισχύσει τις σχέσεις ανάμεσα στην Αφρικανική Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο, εάν μπορεί να στραφεί προς τα εκεί, θα ήταν κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό και μάλιστα στρατηγικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποτελείται ένα από τους κύριους λόγους για τους οποίους θα πρέπει να στηρίξουμε αυτή την ε, ιδέα για αυτό το μέσο. Η άποψή μου αυτή. Βέβαια δεν θα έχει λόγο ύπαρξη όμως, δεν θα στηριχτεί εάν δεν υπάρξει η πολιτική βούληση της Ευρώπης εκεί που χρειάζεται να δράσει στην Αφρική, εκεί που το χρειάζεται όπως στην Σαχέλ όπου απειλείται άμεσα η σταθερότητα και για την ασφάλεια την ευρωπαϊκή όπως και για την Αφρική και υπάρχει τρομερό συμφέρον της Ευρώπης να ενεργήσει κατά όσων μετα... διακινούν ναρκωτικά και πολλούς άλλους ε, ε, με μια σταθερότητα. Είναι προς το συμφέρον μας εκεί να δράσουμε. Χρειάζεται πολιτική βούληση ε, ε, ακριβώς να είμαστε παρόντες ε, και θα πρέπει και η Άστον να το προωθήσει, να είμαστε ακριβώς παρόντες εκεί, να έχουμε ακριβώς μια εικόνα ορατή από όλους εκεί. Σας ευχαριστούμε. Ναι, ο συνάδελφος ζήτησε το λόγο. Ακούστε, θα πρέπει και την υπηρεσία εξωτερικής παρέμβασης να μας βοηθήσει. Κάτι συγκεκριμένο να ρωτήσω. Εδώ πρόκειται για αυτή την εταιρική σχέση με την Αφρικανική ακριβώς Ένωση. Και έχουμε να κάνουμε και με θέματα ασφάλειας. Αν υπάρξει ένα πρόβλημα σε επίπεδο ασφάλειας ε, μετά από μια εκλογή, ας πούμε, αποτυχημένη, είτε με ενωθία στην εκλογή αυτή, τι γίνεται. Θύνεται και θέμα παρέμβασης. Αν αυτό δεν μπορεί να το ρυθμίσει κανείς με εθνικά μέσα, τότε αυτό το θέμα τίθεται. Ποιος θα είναι ο αρμόδιος για να διαρχιστεί στην παρόμοια κρίση για τη στρατηγική απόσμη παρέμβαση ενός ε, ε, κράτους Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, κατά του backbone του, στην ακτή ελεφαντιστή. Τι ακριβώς, ποιος ηγείται υπό την ηγείτα πιανού σε διμερές επίπεδο, το πλαίσιο δεν είναι και το κατάλληλο κατά την άποψή μου γιατί δεν γίνεται από εκεί, δεν υπάρχει συνομιλητής. Άρα λοιπόν είναι υπερεθνικό το πλαίσιο. Υπάρχει μια δυνατότητα από πλευράς Ευρωπαϊκής να παρεμβαίνει σε παρόμοια καταστάσεις, στιγμές και θέματα και σε ποια θεσμικά πλαίσια ακριβώς ε, εντάσσεται εσείς την παρέμβαση, την επέμβαση αυτή. Ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στην ε, Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Δεν ξέρω ποιος την εκπροσωπεί. Δεν έχω το όνομά σας. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω να σχολιάσω ε, γενικότερα πριν απαντήσω την ερώτηση του αξιότιμου ε, βουλευτή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κέντρο Διαχείρισης της Αναπτυξιακής Πολιτικής. Πολύ εύστοχη η ανάλυση τους και περιστατωμένη. Γενικά συμφωνούμε με τα συμπεράσματά τους. Όχι μόνο εκείνοι, αλλά και άλλοι ομιλητές ε, υπογράμμισαν την ευκαιρία που αποτελεί το Παναφρικανικό Πρόγραμμα ενώ ταυτόχρονα μας προειδοποιεί για τους πιθανούς κινδύνους για να χρησιμοποιήσω τη μεταφορά του αυτοκινήτου που αναφέρθηκε. Μπορεί το αυτοκίνητο να μην λειτουργούσε καλά και χρειάζεται αλλαγή κινητήρα. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε πρόσφατα. Ε, αρχίσαμε ένα προβληματισμό, μια περισυλλογή ε, αυτή τη στιγμή στο Συμβούλιο με τα κράτη-μέλη για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις επιδόσεις μας. Διότι ακούσαμε από τον αξιότιμο συνάδελφο από την Αφρικανική Ένωση ότι οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, Αφρικής και η σημασία τους δεν αφισβητείται από κανένα. Αλλά αυτό που δεν έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα να κάνουμε ε, να βρούμε το σωστό μοντέλο ή την κατάλληλη εκείνη φόρμουλα για να υλοποιήσουμε, να εφαρμόσουμε την πολιτική βούληση που υπάρχει εκατέρωθεν. Γι' αυτό εκινήσαμε τούτη εδώ τη διαδικασία συλλογής και δεν μπορεί φυσικά να είναι μονομερής. Χρειάζεται πολύ ισχυρή υποστήριξη και συμμετοχή από τους Αφρικανούς βεβαίω εταίρους, αλλά και από το Κοινοβούλιο σας και από το Παραφρικανικό Κοινοβούλιο και τις οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών. Αυτό προτιθέμεθα και να κάνουμε. Αυτή στιγμή ε, Είμαστε έτοιμοι ε, και έχει επιτευχθεί συνένεση μεταξύ των κρατών μελών για το τι θα προτείνουμε. Χωρίς να σας αποκαλύψω πάρα πολλά, γιατί ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση, στόχος είναι να δρομολογηθεί και να θετεθεί ως προτεραιότητα ό,τι ε, ήταν στα προγράμματα δράσης για τα επόμενα τρία χρόνια. Και εδώ έρχεται και συνδέεται αυτό με το σημερινό. Κρίμα που το χρονοδιάγραμμα μας αναγκάζει να κάνουμε τέτοιες διαπραγματεύσεις ε, παράλληλα, ε, γιατί δεν μπορούμε να συζητήσουμε μία συζήτηση για τα χρηματοοικονομικά, ενώ ταυτόχρονα, όπως εξηγήθηκε πολλές φορές σήμερα, τέλη του 2013, αρχές του 2014, θα έχουμε σύνοδο κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικής. Λοιπόν, Οπωσδήποτε ένας από τους τομείς που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι η ανάγκη να ενισχυθεί ο πολιτικός διάλογος. Άκουσα μια έκκληση, ίσως και ένα παράπονο, να εκφράζει ο κύριος Μπέρμαν, ότι θα πρέπει κάθε Άστο να είναι πιο παρούσα. Θα της το διαβιβάσω. Είμαι σίγουρος ότι έχει την πρόθεση αυτή. Δεν χρειάζεται να μπω σε λεπτομέρειες της δυσκολίας ε, του έργου της για να το καταλάβει. Δεν μπορεί να είναι πανταχού παρούσα. Δεν ε, διαμαρτύρονται και παραπονιούνται μόνο οι Αφρικανοί αλλά και άλλοι. Αφήστε δε που έχει πάει ήδη μερικές φορές στην Αφρική. Αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε να επανεκκινήσουμε τον ε, διάλογο σε υπουργικό επίπεδο και να έχουμε και πιο τομεακούς διαλόγους για να μπορούν ε, οι επίτροποι και οι υπουργοί. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν ε, πολλές συναντήσεις ομολόγων και το Κολεγίου των Επιτρόπων, του Σώματος των Επιτρόπων και άλλες επαφές ε, ουσιαστικά σε καθημερινή βάση μεταξύ των δύο επίρων και των όσων προσπαθούν να λύσουν κοινά προβλήματα όπως προηγουμένως ακούστηκε. Απαντώ σε ορισμένα από τα ερωτήματα που ετέθησαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Πρώτο αυτό το ζήτημα του κοτονού. Συγγνώμη, λέει η πρόεδρος, ε, δεν έχουμε χρόνο, θα θέλατε να ολοκληρώσετε. Καλώς. Τότε να απαντήσω την ειδική ερώτηση που έκανε ο κύριος Γκέρενς. Πρέπει να σας πω ότι οι δικές μας προσπάθειες πηγαίνουν στην τελείως αντίθετη κατεύθυνση. Οι κρίση στην Αφρική θα πρέπει να επιλύονται από τους ίδιους τους Αφρικανούς. Αυτό είναι το πρόβλημα του, ότι δεν έχουν κάνει κτήμα τους αυτό το θέμα. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε ε, στην εταιρική σχέση ειρήνης και ασφάλειας, να μπορούν να έχουν σε επιφυλακή στρατεύματα αφρικανικά που να μπορούν να ε, αναπτύσσονται σε σύντομο χρονικό διάστημα όπως ε, ε, ήταν το θέμα της ακτής ελεφαντοστούν. Οι Αφρικανοί έχουν ένα ωραίο πλαίσιο για το πώς θα λειτουργούν όταν έχουμε αντισυνταγματικές αλλαγές καθεστώτων και κυβερνήσεων αλλά χρειάζεται λίγο να ενδυναμωθεί αυτό ως μηχανισμός και αν γίνεται να επεκταθεί και να γίνει ένα παναφρικανικό πρόγραμμα, εάν εγκριθεί. Ευχαριστώ. Merci beaucoup. Je donne maintenant la parole ευχαριστώ. Οι εμπειρογνώμονες έχουν τώρα το λόγο. Για τρία λεπτά παρακαλώ ο καθένας. Um, thank you very much. Uh, ευχαριστώ πολύ. Θα... Σε σχέση με τα θέματα που ήδη αναφέραμε, πιστεύω ότι αντιλαμβανόμαστε αρκετά ξεκάθαρα τους κινδύνους και τις ευκαιρίες του Παναφρικανικού Προγράμματος από την πλευρά μας στο κέντρο του ECTPM θεωρούμε ότι είναι μια εξαιρετική ευκαιρία αλλά μόνο εφόσον αντιμετωπιστούν οι κρίσιμοι κίνδυνοι που τους συνοδεύουν. Χρειάζεται λοιπόν να ληφθούν μια σειρά συμπληρωματικών μέτρων γιατί το Παναφρικανικό Πρόγραμμα δεν θα λύσει όλα τα προβλήματα, δεν μπορεί η χρηματοδότηση να αντικαταστήσει έναν διάλογο ο οποίος πρέπει να διεξαχθεί σε παναφρικανικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο. Και από αυτό το πρίσμα, ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα είναι ο ρόλος του Κοινοβουλίου εδώ, αλλά και ο ρόλος του Παναφρικανικού Κοινοβουλίου. Να τρόπους στο πλαίσιο των κανονισμών στους οποίους λειτουργείται έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι το πρόγραμμα θα γίνει κτήμα των Αφρικανών και θα είναι αποτελεσματικό και από την πλευρά των άσκησης πολιτικής στην Αφρική και από την πλευρά της Ευρώπης. Το πρόγραμμα αλλά και η κοινή στρατηγική πρέπει να έχουν απτά αποτελέσματα και να σημαντικά αποτελέσματα στην, επιτόπου στην Αφρική. Στο πλαίσιο του Παναφρικανικού προγράμματος θα πρέπει οι πολίτες οι Αφρικανοί να έχουν, ε, την, να έχουν λόγο στον τρόπο με τον οποίο υλοποιείται το πρόγραμμα και να έχουν την εποπτεία του. Σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ και που σεβαστήκατε και το χρόνο. Θα δώσω το λόγο για τρία λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν μίλησα για τους κινδύνους. Αυτό το πρόγραμμα δεν έχει κανένα κίνδυνο, διατρέχει κανένα κίνδυνο. Στο ίδιο μήκο κύματο με την Επιτροπή και με την Υπηρεσία Εξωτερική Δράση. Άρα λοιπόν είμαστε υπέρ τη πρόταση. Αυτό ζητούσαμε πάντα άλλωστε. η κοινή στρατηγική δεν εφαρμόζεται ιδιαίτερα επειδή δεν υπάρχει ένα ειδικό μέσο με τα απαραίτητα μέσα που να διαθέτει και γι' αυτό το παναφρικανικό πρόγραμμα θα είναι όμως μια προστιθέμενη αξία για την εταιρική αυτή σχέση. Το όλο πλαίσιο πάντως είναι μια βελτίωση και αυτό για να ισχύσουν όλα αυτά για τη συνθήκη για την Αφρική που να αντιμετωπίσει την Αφρική σαν μια ενότητα σχετικά με την ειρήνη και στην ασφάλεια αυτά που ρωτήθηκαν. Το μέσο αυτό αποτελεί το τέλειο παράδειγμα της προστιθέμενης αξίας της εταιρική σχέσης. Αυτό δίνει αυτά αποτελέσματα, συνεχίζει να δίνει, γιατί έτσι η αρχιτεκτονική αυτή αφρικανική μπαίνει σε κατάλληλα πλαίσια και για να ανταποκριθούμε σε αυτές τις προκλήσεις ε, υπάρχει μια λύση που μπορεί να είναι στη ρίζα του να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, στην ανάπτυξη δηλαδή και το μέσο αυτό αποτελεί άριστο παράδειγμα γιατί για την απασχόληση και θα μπορέσει να ισχύσει και να δώσει απάντηση σε αυτά τα προβλήματα. Αυτή η εταιρική σχέση είναι ειδική σε αρκετές πτυχές της. Αυτό που σήμερα συμβαίνει στην Αφρική και στην ε, Ευρώπη, στην Ευρώπη επηρεάζει την Αφρική και αυτό που έχει να κάνει με την Αφρική επηρεάζει την Ευρώπη κυρίως. Αλλά και με τις αραβικές χώρες το ίδιο. Είμαστε οι φυσικοί εταίροι και είτε θα πετύχουμε από εκείνο, είτε θα αποτύχουμε όλοι μας. Και αυτό το μέσο δεν είναι πανάκια, αλλά σίγουρα θα βοηθήσει για την πραγματική εφαρμογή του σχεδίου δράσης αυτού, για αυτή την κοινή στρατηγική. Σας ευχαριστώ, λέει Πρόεδρο, σας ευχαριστώ για τη συζήτησή μας, που σίγουρα θα μας εμπνεύσει για τις τροπολογίες μας για την πολιτική αυτή ανάπτυξη. Και και τώρα τα σημεία 18 και 19 της ημερησίας διάταξης, με αυτά θα ασχοληθούμε, κανόνες και διάδοση του προγράμματος πλαίσιο ερεύνας και καινοτομίας ορίζον 2020, κανόνες διάδοσης των αποτελεσμάτων και θέσπιση του προγράμματος πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία ορίζον 2020. Πρόκειται για δύο γνωμοδοτήσεις ο κύριος Μπιλ Νιούτον Ντάν είναι ο συντάκτης τους. Γνωμοδοτήσεις για την Ήτρε. Έχουμε το πρώτο σημείο, το 18, με ένα ενιαίο πρόγραμμα πλαίσιο στήριξης της έρευνας και της ονοτομίας για την περίοδο 2014-2020 Επίση θα δούμε και τις κανόνες συμμετοχής σε αυτό το πρόγραμμα. Μετά δε, δεν χρειάζεται τώρα να σας πενθυμίσω ότι το όνομα της Επιτροπής βασίζεται σε τρεις και σε τρία και συστατικά την αριστεία σε επιστημονική βάση, μια leadership βιομηχανική και τα πλαίσια για τον ανταγωνισμό και την απάντηση στα στις προκλήσεις και αυτό δείχνει και την φιλοδοξία αυτού του ε, προγράμματος πλαισίου να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε, να δώσουμε μια απάντηση σε αυτές τις προκλήσεις. Δεν θα χάνουμε χρόνο, αλλά ο κύριος Νιούτον Ντάν έχει το λόγο για να μας πει πώς έχουν τα πράγματα με αυτές τις δύο γνωμοδοτήσεις του. Έχετε το λόγο κύριε Νιούτον Ντάν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε είπατε πολλά και αυτό με διευκολύνει. Λοιπόν, υπάρχουν δύο σημεία στην ημερήσια διάταξη, το 18 και τα 19, τα οποία τα εξετάζουμε από κοινού, γιατί και τα δύο αφορούν στο πρόγραμμα Horizon 2020. Το σημείο 18 αφορά στις κανόνες και τη διάδοση, ενώ το 19 είναι η θέσπιση του προγράμματος. Η γραμματεία, με την σοφία που τη χαρακτηρίζει, προτείνει ως ε, προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών τις 12 Ιουλίου την ώρα του μεσημεριανού φαγητού, στις 12. Επομένως, ε, αν και δεν είναι όλοι παρόντες, θα σας ζητήσω την προσοχή σας, έτσι ώστε να καταλάβουμε εάν υπάρχουν ε, τροπολογίες και να, αν πρόκειται η Επιτροπή να αλλάξει πολύ το, τη γνωμοδότηση. Για το πρόγραμμα Horizon, 12 επιτροπές του Κοινοβουλίου θα διατυπώσουν γνωμοδότηση. Επομένω πρέπει να είμαστε πολύ σαφείς. Και έχουν πάντα πολύ αυστηρές προθεσμίες για την κατάθεση του, των τροπολογιών. Με ανησυχεί λίγα και αυτό και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Τώρα όσον αφορά το σημείο 19, η πρόταση της Επιτροπής χωρίζεται σε τρεις πυλώνες, την ε, ε αριστεία, την καινοτομία και τις κοινωνικές προκλήσεις. θεωρώ ότι από την πλευρά μας εμείς θα πρέπει να εστιάσουμε στις παγκόσμιες προκλήσεις που προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε. Για παράδειγμα, την επιστηστική ασφάλεια, την υγεία και την κλιματική αλλαγή, δηλαδή όλα αυτά τα μεγάλα πράγματα που βλέπουμε να έρχονται και πρέπει να βρούμε καλύτερες λύσεις από τις σημερινές. Λοιπόν, ε, προτείνω στους συναδέλφους να εστιάσουν σε του σε αυτόν τον τομέα στις τροπολογίες τους. Νομίζω ότι αυτό είναι ο τομέα στον οποίο η δικιά μα επιτροπή μπορεί περισσότερο να συνεισφέρει σε σχέση με τι υπόλοιπε 11. Εξίσου σημαντικό είναι οι κανόνε που, που καθορίζουν ποιο μπορεί να συμμετάσχει στο Horizon 2020. 2020. Ε, Προτείνω μια σειρά τροπολογιών έτσι ώστε να διασφαλιστεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή στο πρόγραμμα και μια όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας που θα γίνουν στο πλαίσιο του Horizon 2020. Γνωρίζουμε, για παράδειγμα, στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής χρειάζεται να υπάρξει μεταφορά τεχνογνωσίας προς τις λιγότερο αναπτυγμένε χώρες Ή να, αυξηθεί, αυξηθούν οι συμπράξεις ιδιωτικού δημόσιου τομέα. Θα ήμουν λοιπόν ευτυχής εάν και άλλοι συνάδελφοι προτείνουν τροπολογίε επί των ζητημάτων αυτών, συμπεριλαμβανομένων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Υπάρχει λοιπόν ένα ζήτημα το οποίο με απασχολεί ιδιαίτερα, ότι θα δαπανηθούν πολλά χρήματα για την υγεία τα επόμενα χρόνια, γιατί μια και αυξάνεται ο πληθυσμό τη γης ε, η υγεία είναι σημαντικό πρόβλημα, αλλά σε συνδυασμό με την κλιματική αλλαγή, σε συνδυασμό με την μετανάστευση, γίνεται ακόμα πιο ε, δύσκολο πρόβλημα. Και γι' αυτό πρέπει, πιστεύω, να πιέσουμε την Επιτροπή να αφιερώσει όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο μπορεί σε αυτό το θέμα. Μια και λοιπόν έχουμε λίγο χρόνο στη διάθεσή μα για να καταθέσουμε τροπολογίε, σε αυτού του τομεί θέλω να προτείνω να εστιάσουμε. Σα ευχαριστώ, κυρία Κέλλερ. Με μεγάλη χαρά σας ξαναβλέπω στην Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ε, από πλευρά Πρασίνων είμαι σκιώδη εισηγήτρια εγώ. Ε, ευχαριστώ πολύ για την εξαιρετική σα έκθεση. Μπορούμε να την υποστηρίξουμε πλήρω εδώ στην Επιτροπή μα. Δεν χρειάζεται να τονίσω ότι για να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή θα πρέπει ε, οι αναπτυσσόμενες χώρες να προχωρήσουν, να ξεφύγουν από μια κοινωνία με ε, εντατική παραγωγή ε, διοξιδίου του άνθρακα και να πάνε σε μια άλλη ανάπτυξη. Και πολύ σημαντικό αυτό που είπατε για την ιατρική. Τεχνολογία καινοτομία θα πρέπει να μας βοηθήσει και να μεταφέρουμε την τεχνογνωσία αυτή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Διεθνής Κοινότητα, πώς να το πω, έχει συμφωνήσει ήδη για τη μεταφορά τεχνογνωσίας, αναφέρεται και συμφωνία TRIPS για τα πνευματικά δικαιώματα, ε, για ε, τις συμβάσεις για το κλίμα, παντού αναφέρεται. Η μεταφορά της τεχνογνωσίας αυτή καθ' αυτή είναι κάτι το οποίο έχει δεχθεί η διεθνή κοινότητα, αλλά πολύ συχνά λείπουν οι συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς θα υλοποιηθεί αυτή η καλή πρόθεση. Δεν εφαρμόζονται αυτά. Και πιστεύω ότι ο Horizon 2020 θα είναι η κατεξοχήν ευκαιρία να ε, γίνει πράξη αυτή η πρόθεσή μας. Και ελπίζω οι τροπολογίες της Επιτροπής ΔΕΒΕ να γίνουν δεκτές από την Επιτροπή Βιομηχανίας, Ήτρε. Καλωσορίζω τη γνωμοδότηση και την έκθεση για τη συνεργασία με τις αναπτυσσόμενες χώρες για την έρευνα. Θα κάνουμε μέχρι την Πέμπτη λίγες τροπολογίες, αλλά προς αυτή ακριβώς την κατεύθυνση. Υποστηρίζω απολύτως την πρότασή σας. Έχουμε συγκεκριμένα παραδείγματα όπως ένα πουλ για ε, ε, διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή να διευκολύνεται η αδειοδότηση σε τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Συγκεκριμένες προτάσεις θα κάνουμε λοιπόν έτσι ώστε να εμπλουτίσουμε την έκθεσή σας λίγο. Ζητώ συγγνώμη, πρέπει να φύγω γιατί συζητούμε τον προπολογισμό στην άλλη μου επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Κέλλερ. Και θα δώσω τώρα το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που εκπροσωπείται από τον κύριο Τζον Κλάκστον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, καλωσορίζουμε τη συζήτηση στην Επιτροπή σας και το ενδιαφέρον που δίδεται για τη διεθνή διάσταση της κοινωνικής καινοτομίας ε, και γενικά ε, θυμίζουμε ότι η διεθνή συνεργασία είναι σημαντική διάσταση του ορίζοντα 2020, πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία που έχει βασικό στόχο ακριβώς τη βοήθεια να δοθεί ανάπτυξη ευφυής, ε, βιώσιμη και γένεια ώστε ω τμήμα τη στρατηγικής για το 2020. Συμφωνούμε με τις απόψει που εκφράστηκαν στην ανάλυση τη επιτροπή σα. Ωστόσο θα θέλαμε να θυμίσουμε ότι ο ορίζουν 2020 δίδει ένα πλαίσιο μέσα στο το οποίο μπορούν να αναπτυχθούν λεπτομέρειες. Και υποστηρίζουμε και σημειώνουμε ότι ορισμένα από τα ειδικά σχόλια των τροπολογιών για τις κοινωνικές προκλήσεις έχουν ήδη αναφερθεί. Ας πούμε η διεθνή συνεργασία και όλα αυτά αναφέρονται σε ένα ειδικό πρόγραμμα που είναι τμήμα του πακέτου του Horizon 2020. Παράδειγμα. τομεακή ε, διεθνή συνεργασία. Ε, υπάρχει ένα τμήμα για τη βοήθεια σε αναπτυσσόμενες χώρες με συγκεκριμένα ε, παραδείγματα των τομέων και των κλάδων που θα μπορούσαν. Ας πούμε κλινικές δοκιμές, εταιρική σχέση, αυτό για την έρευνα στα σπάνια νοσήματα και η υπόθεση του διακρατικού διακυβερνητικού πάνελ για την κλιματική αλλαγή. Σημειώνουμε αυτά που λέτε για τη δωρεάν πρόσβαση, ο access και ε, ο Horizon 2020 θα βασιστεί σε ένα τέτοιο πιλωτικό πρόγραμμα του προγράμματος πλαίσιο 7 για την έρευνα. Ό,τι αφορά τις επιστημονικές δημοσιεύσεις επίσης ε, θα είναι ανοιχτή και δωρεάν η πρόσβαση δηλαδή και στα δεδομένα της έρευνας και για τα δεδομένα θα πρέπει να θυμίσουμε ότι η πρόσβαση δεν θα πρέπει να υπονομεύει τη συμμετοχή ε, εταιριών και ε, μικρομεσαίων. Γι' αυτό υπάρχει ένα μέλημα θεμητό για την προστασία των εμπορικών συμφερόντων και της πνευματικής ιδιοκτησίας και των πνευματικών δικαιωμάτων. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να δημοσιεύσει μια ανακοίνωση για τη διεθνή συνεργασία στην έρευνα και την καινοτομία και μεταξύ άλλων θα ασχοληθεί με τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας για την ανάπτυξη και πώς μπορεί αυτό να ενταχθεί στην έρευνα και στην καινοτομία και στις αντίστοιχε πολιτικές. Το Σεπτέμβριο προτιθέμεθα να δημοσιεύσουμε αυτή την ανακοίνωση. Και με την άδειά σας να δώσω το λόγο στον συνάδελφο κύριο Σούλτ που θα σας πει τα νομικά ζητήματα. Μια μικρή λεπτομέρεια. Σημειώσαμε ότι σε ό,τι αφορά τους κανόνες συμμετοχής Υπάρχει ε, μια συγκεκριμένη διατύπωση για τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, δημοσίου και με δημόσιο τομέα. Είναι πάρα πολύ τεχνική αυτή η διαδικασία. Ε, Δεν θα πρέπει όμως αυτό να εγγραφεί στους κανόνες ε, συμμετοχής, αλλά στο πλαίσιο, τον κανονισμό πλαίσιο για τον ορίζοντα 2020. Είναι πάρα πολύ τεχνικό όμω αυτό το θέμα και μπορεί ε, να εξηγηθεί αν θέλετε διμερώς να σα δώσουμε περισσότερες εξηγήσει. Ευχαριστώ πολύ. Θα ξαναδώσω το λόγο στον κύριο Νιούτον Ντάν για να ολοκληρώσει. Well, thank you very much. We, we seem to... Ευχαριστώ λοιπόν. Φαίνεται πως συμφωνούμε γενικά και αυτό είναι πολύ καλό. Θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό το πολύ τεχνικό ζήτημα που έθεσε ο τελευταίος ομιλητής από την Κομισιόν. Μήπως θα μπορούσατε να μου στείλετε ένα email που να, μας, να μου εξηγείτε πού είναι το τεχνικό πρόβλημα και τι πρέπει να γίνει τελικά. Ε, γιατί ίσως εμείς στην, στην Επιτροπή να μην καταλαβαίνουμε την τεχνική αυτή λεπτομέρεια, αλλά να μπορέσουμε να την εξηγήσουμε σε όλους τους άλλους. Αν μπορείτε να μου το στείλετε αυτό θα ήμουν ευγνώμων. Ευχαριστώ. Να σας υπενθυμίσω κάτι ότι 12 Ιουλίου το μεσημέρι είναι προθεσμία για τις τροπολογίες και ότι αυτό θα το ψηφίσουμε στην πρώτη μας συνάντηση στις 3 Σεπτεμβρίου. Πάμε παρακάτω. Το σημείο 20 της ημερήσιας διάταξης. Ανταλλαγή απόψεων για το σχέδιο έκθεσης για τις εργασίες της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης ή εκπροσώπησης ΑΚΕ Ευρωπαϊκής Ένωσης ο κύριος Νόρμπερτ Νόιζερ είναι ο συντάκτης ε, αυτής της έκθεσης. Είναι η ετήσια έκθεση υπό τον κύριο Νόρμπερτ Νόιζερ, μέλος ε, της ε, κοινοβουλικής αυτής συνέλευσης, η οποία το 2011 συνέχισε με τις τακτικές εργασίες με δύο ολομέλειες και με τις μόνιμες αντιπροσωπείες που συνεδρίασαν. Δυστυχώς, δυστυχώς όμως η συμμετοχή Ευρωπαίων μελών συναντήσει αυτές μειώθηκε η συμμετοχή τους ε, και υπήρξε μια ιδιαίτερη κριτική που ασκήθηκε από τα μέλη όπως και τη γραμματεία και ο κύριος Νόρμπερ Νόιστερ θα λάβει το λόγο για να μας ε, παρουσιάσει την εκθεσή του. Ja, vielen Dank, Frau. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σήμερα Έχουμε την έκθεση για τα πεπραγμένα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ε, ΑΚΕ Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η πρώτη μας συζήτηση, χωρίς έγγραφο προς το παρόν. Η δεύτερη συζήτησή μας θα ακολουθήσει αμέσως μετά τις θερινές διακοπές της 3 Σεπτεμβρίου και η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών είναι η επόμενη ημέρα, 4 Σεπτεμβρίου. Οπότε αν έχουμε τροπολογίες αμέσως μετά τις διακοπές θα πρέπει να στρωθούμε στη δουλειά. Όπως είπατε και εσείς πέρυσι, η ε, συνέλευση της εκπροσώπηση συνεδρίασε δύο φορές. Πέρσι το Μάιο στη Βουδαπέστη ήταν η πρώτη και η δεύτερη συνεδρίαση τον Νοέμβριο του 2011 στη Λομέ του Τογκό. Έχουμε δέκα ψηφίματα συνολικά εγκρίνει και δύο δηλώσεις και επιπλέον το Προεδρείο ε, ΑΚΕ Ευρωπαϊκής Ένωσης έστειλε εξεταστική των πραγμάτων αποστολή στον Ανατολικό Τιμό. Η ε, Επίτροπος μας, η Επίτροπη μας και ε, για την πολιτική, την αναπτυξιακή. Εργάζονται πολύ ε, σε αυτή την κατεύθυνση. Ο κύριος Πίμβαλξ ήταν παρόν σε όλες τις ε, συνελεύσεις ομερούς. Αυτό θα ήταν καλό και για την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Θα αναβαθμιζόταν πάρα πολύ η συνέλευση της εκπροσώπησης αν ερχόταν κάποια φορά η κυρία Άστον. Κυρία Πρόεδρε, σωστά επιπλήξατε, επισημάνατε ότι στις Βρυξέλλες ε, ή στην Ευρώπη όταν έρχονται ε, οι ΑΚΕ δεν παρευρίσκονται πολλοί βουλευτές ε, και αυτό μας το προσάπτουν. Ναι, αλλά όταν συνεδριάζει εδώ η Σομερίσα και η Ευρωπαϊκή Ένωση, γίνεται παράλληλα με άλλε συνεδριάσει που προσκρούν στη συνεδρίαση αυτή. Και αυτό το χρησιμοποίησαμε ω ε, αφορμή από την επόμενη φορά, από το Σεπτέμβριο, να αλλάξουμε το σύστημα και να ε, ορίζουμε τι συνεδριάσει την Πέμπτη και την Παρασκευή. Έτσι ώστε τουλάχιστον την Πέμπτη το απόγευμα και την Παρασκευή να μην έχουμε άλλε επιτροπέ ε, που να συνεδριάζουν παράλληλα και να δούμε πώ θα έχει προσέλευση από εκεί και πέρα. Και μήπως αυξηθεί η συμμετοχή των Ευρωβουλευτών. Πέρυσι η ομάδα εργασίας ασχολήθηκε με τις ομάδες εργασίας της ε, συνέλευσης εκπροσώπησης, ολοκλώρισε το έργο της. Η ομάδα εργασίας είχε συσταθεί για να εκτιμήσει τον πολιτικό ρόλο και Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τον ενισχύσει και η διαδικασία να διαμορφωθεί πιο αποτελεσματικά δεν μπόρεσαν να εφαρμοστούν ήδη από το 2011 όλες οι προτάσεις που κάναμε για τη μέθοδο εργασίας, οπότε έχει απομείνει αρκετή δουλειά και για φέτος. Τα διάφορα ψηφίσματα που εγκρίναμε, δεν θέλω να σας τα αναφέρω λεπτομερώς, πιστεύω ότι είναι πιο σημαντικό να καταλάβουμε ποια είναι η φιλοσοφία που διέπει τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρών ΑΚΕ. Γιατί αυτή η ισομερή συνελευσή είναι πολύ σημαντικός διάλογος βορρά-νότου. Εάν δω το παράδειγμα των ΕΠΑ, των ε, εμπορικών αυτών συμφωνιών, για να μπορέσουμε να έχουμε και κοινέ ε, συμφωνίες. Επίσης σημαντικό είναι η κοινωνία των πολιτών σε βορρά και νότο να συμμετέχει και να ακούγονται και τα τοπικά προβλήματα καλύτερα στις ισομερείς. ΑΚΕ. Επίσης είναι πολύ καλή η συνεργασία και ο διάλογο αυτό με τους βουλευτέ, όχι μόνο για να καταλήγουμε σε κοινέ θέσει. Παράδειγμα, η Αραβική Άνοιξη το 2011 ε, συζητήθηκε ε, εκτενέστατα και στις δύο συνεδριάσεις. Ακόμα και αν έχουμε μεγάλες διαφορές στην αντίληψή μας με τις χώρες ε, και είναι καλό να έχουμε αυτές τις ανταλλαγές απόψεων, είτε τις επίσημες είτε τις άτυπες. Και για μένα δεν είναι ίσονο σημασία ε, οι βουλευτές ΑΚΕ ε, να εργάζονται με δημοκρατικές αρχές ε, και μάλιστα αυστηρά δημοκρατικές αρχές και εμείς όταν πρόκειται για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πραξικοπήματα σε χώρες και τα αναφέρουμε και τα καταδικάζουμε από κοινού. Είναι μεγάλη δημοκρατική ακτινοβολία της ΑΚΕ Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις δικές μας αξίες και αρχές. Να σας πω με τι ασχοληθήκαμε. Υποστήριξη από τον προπολογισμό, προβλήμα της ακτή ε, ελεφαντοστού, ε, ρήπαση του νερού, καταπολέμηση του AIDS, ε, το θέμα των χρεών επίσης. Το θέμα των ατόμων με αναπηρία στις αναπτυσσόμενες χώρες και τα προβλήματα στο κέρα της Αφρικής και ιδιαίτερα η κατάσταση ασφαλείας στη Σομαλία, καθώς επίσης και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ερυθρέα. Ευχαριστώ. Merci. Ευχαριστώ. Και τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ζωσά, το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρόκειται για μία ανταλλαγή απόψεων. Τον κύριο Νόιζα λοιπόν θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για όσα είπε ε, για τον Επίτροπο, τον Αρμόδιο που ιδιαίτερα προσέχει αυτό τον απασχολεί ιδιαίτερα και προσπαθεί να συμμετέχει σε όλες τις συναντήσεις αυτής της ε, Σοβαρής Επιτροπής. Θεωρεί ότι είναι μια κάποια στιγμή σημαντική όπου οι δημοκρατικές αρχές ε, συναντούνται το χρόνο και, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έκθεση τώρα. Έχουμε τις δραστηριότητες ε, που έχουν σημειωθεί και πολύ σημαντικά που έχει στο παρελθόν ακριβώς θα έχουμε ένα τμήμα που θα έχει να κάνει με την ε, μελλοντική ανάπτυξη. Για αυτή λοιπόν την πτυχή προς τα εκεί θα πρέπει να επικεντρώσουμε την ε, προσοχή μας εδώ στο Κοινοβούλιο. Πολλά νέα σημεία όσο αφορά τη μεθοδολογία, της εργασίας κλπ. Σημαντικό θα ήταν εδώ σε αυτή τη συνέλευση να προσπαθήσουμε να δούμε ποιες είναι οι κοινέ προκλήσεις που απασχολούν όλους για μια πιο σημαντική πολιτική διάσταση να δούμε τι ακριβώς είναι εκεί και ποιες θα μπορούσαν να είναι οι κοινέ λύσεις ε, πάνω σε θέματα και σε προβλήματα που να είναι και γενικότερες σφαιρικές προκλήσεις και μόνο, όχι μόνο προβλήματα των χωρών ΑΚΕ, είτε προβλήματα που μπορεί να ρυθμίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις σχέσεις της απευθείας με τις χώρες της Αφρικανικής στα Αφρικής, θέματα όπως οι κλιματικές αλλαγές, ε, μεγάλες ε, συναντήσεις ε, και τα επόμενα χρόνια θα έχουμε μια αναθεώρηση σε παρόμοια θέματα, να δούμε και στον μέθνενή τι γίνεται με το 2015, με την ασκούμενη πολιτική για τους ε, για την έκθεση επίσης για τον ρόλο των χωρών στα πλαίσια της συμφωνίας Λισαβόνας, ε, αλλά ίσως θα ήταν και η κατάλληλη στιγμή να δούμε το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στις χώρες ΑΚΕ. Η δικά της δυνατότητα συγκενώνεται γύρω από τις Βρυξέλλες και δεν προχωράει παραπέρα. Η σχέση με τον Χορονακέ και με την ομάδα των 77 και οι χώρες ΑΚΕ στις διεθνείς διαπραγματεύσεις πώς επηρεάζουν την πραγματικότητα και να ξεπεράσουν αυτό το σχεδιασμό με ιδιαίτερο προσανατολισμό που συγκεντρώνεται ας πούμε στις συναντήσεις και στα όσα έχουν να κάνουν με την απόφαση του Κοτονού και να πάνε προς κάτι το σφαιρικότερο. Αυτή είναι και η πρώτη σκέψη, ο πρώτος συλλογισμός της Επιτροπής για να βοηθήσουμε στη σχετική συζήτηση και το 2011 είχαμε σημαντικότατα ψηφίσματα και οι προοπτικές το όραμα για το μέλλον αυτό θα πρέπει να αναπτυχθεί περισσότερο και να αποτελέσει αίτιο για να ε, ενδιαφερθούν ακόμα περισσότερο οι βουλευτές για να συμμετάσχουν γιατί ε, έχει δίκιο η πρόεδρος που εξέφρασε τη λύπη της γιατί δεν συμμετέχουν πολύ όπως και η επέναντι πλευρά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε λέει η πρόεδρος. Κανείς άλλος δεν έχει ζητήσει το λόγο και πάλι ο κύριος δεν έχει το λόγο, όχι. Ολοκληρώσαμε λοιπόν την πρώτη ανταλλαγή απόψεων και τις τροπολογίες σας μπορείτε να τις καταθέσετε μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου το μεσημέρι. Τις 10 του μήνα θα ψηφίσουμε. Ε, Έχουμε το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη που είναι ανταλλαγή απόψεων ε, με την κυρία Κοζάκου Μαρκούλη έρατο στις 5 όμως ε, και λείπουν λοιπόν, 7-8 ε, λεπτά, 10 λεπτά και διακόπτουμε λοιπόν την συνεδρίασή μας για 10 λεπτά για να έρθει η Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου. Ευχαριστούμε. Αν θέλετε να καθίσετε παρακαλώ για να επαναληφθεί η συνεδρίαση της Επιτροπής μας μετά το διάλειμμα. Θα θέλαμε να σας πούμε ότι έχουμε τη χαρά να ε, υποδεχόμαστε την κυρία ε, δόκτωρα Ερατό Κοζάκου Μαρκουλή που είναι Υπουργό Εξωτερικών τη Κυπριακή Δημοκρατία, και θα μα παρουσιάσει τι προτεραιότητε τη Κυπριακή Προεδρία στον τομέα τη ανθρωπιστική βοήθεια. Καταρχάς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε αγαπητή κυρία Υπουργέ για την προθυμία σας να έρθετε στην Επιτροπή μας. Χαιρόμαστε ήδη για την εξαιρετική συνεργασία που ήδη έχουμε αρχίσει το τελευταίο διάστημα, μήνες και εβδομάδες με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Κυπριακή Προεδρία και εγγράφεται πλήρως ε, στο νομοθετικό πλαίσιο και διοργανικό που ετέθησε ισχύ με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας υπάρχουν πολλές προκλήσεις, πολύ συγκεκριμένες τους επόμενους μήνες ε, από την έγκριση της Σύμβασης για την ανθρωπιστική, ε, επισητιστική μάλλον βοήθεια, μέχρι τις διαπραγματεύσεις για το νομοθετικό πλαίσιο, για το μελλοντικό εθελοντικό ε, σώμα για την ανθρωπιστική βοήθεια και το μηχανισμό πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης θα ακούσουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τη σκέψη σας για την πολιτική και ανθρωπιστική κρίση που αντιμετωπίζει σήμερα η Συρία. Είναι ένας πάρα πολύ κοντινός γείτονας της χώρας σας. Ε, υπογραμμίζω ότι η ανταλλαγή απόψεών μας αφορά αποκλειστικά τον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας στα πλαίσια της περιτροπής προεδρίας ε, του Συμβουλίου της Ένωσης. Οποιοδήποτε θέμα που έχει να κάνει γενικότερα με τη συνεργασία, την αναπτυξιακή, μπορεί να τεθεί είτε κατά τη διάρκεια του διαρθρωμένου διαλόγου με τον Επίτροπο Πίμπαλξ, είτε κατά τη διάρκεια της ετήσιας ανταλλαγής απόψεων με την κυρία Άστον, την ύπατη εκπρόσωπο της Ένωσης για τα εξωτερικά θέματα και την πολιτική ασφάλεια και Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κυρία Υπουργέ, με χαρά θα σας δώσω το λόγο για 20 λεπτά περίπου. Παρακαλώ. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής, κυρίες και κύριοι. Είμαι ιδιαίτερος ευτυχής και είναι πράγματι μεγάλη τιμή για εμένα να έχω την ευκαιρία να απευθυνθώ στην Επιτροπή σας και να συζητήσω μαζί σας για αυτό το εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα της ανθρωπιστικής βοήθειας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο τα θεσμικά όργανα όσο και τα κράτη-μέλη, είναι ο μεγαλύτερος δωρητής βοήθειας παγκοσμίω στην αναπτυξιακή συνεργασία και στην ανθρωπιστική βοήθεια. Η Κύπρος είναι ένα νέο μέλος στην οικογένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η συνεισφορά της ως δωρητής είναι σχετικά μικρή. Μιας και στο όχι και τόσο μακρινό παρελθόν η Κύπρος αποτέλεσε χώρα η οποία δέχθηκε βοήθεια και έτσι μπορούμε να αναγνωρίσουμε τη σημασία της ανθρωπιστικής ε, και αναπτυξιακής βοήθειας. Η Κύπρος αναλαμβάνει την προεδρία σε μια δύσκολη συγκυρία Τη στιγμή που οι προϋπολογισμοί για ε, την αναπτυξιακή βοήθεια και για την ανθρωπιστική βοήθεια των κρατών μελών περικόπτονται εξαιτίας της πίεσης από την παγκόσμια οικονομική κρίση. Παρ' όλα αυτά θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διατηρήσει και να ενισχύσει τον ηγετικό της ρόλο στην αντιμετώπιση των πολλαπλών ανθρωπιστικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε αποτελεί πρόκληση για την Κύπρο η ε, συνέχιση του έργου της Δανεικής Προεδρίας. Θα ήθελα προσωπικά να συγχαρώ τους ε, ε, ομολόγους μου και τους συναδέλφους από την Δανία για τον υπαδογματικό τρόπο που επιτέλεσαν το έργο τους καθ' όλη τη διάρκεια της Δανικής Προεδρίας, αλλά και ιδιαίτερα στον τομέα της αναπτυξιακής συνεργασίας και της ανθρωπιστικής βοήθειας. Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να συνεχίσουμε το σημαντικό έργο που ξεκίνησαν σε αυτόν τον τομέα θα ήθελα να σας δώσω μια γενική παρουσίαση των προτεραιοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας. Μετά θα ήθελα να εστιάσω σε δύο συγκεκριμένες ανθρωπιστικές προκλήσεις στην Αφρική, τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνεχίσει να αντιμετωπίζει, δηλαδή τις προκλήσεις στο Σαχέλ και στο κέρας της Αφρικής. στο πλαίσιο αυτό η Κυπριακή Προεδρία θα εστιάσει στα εξής ε, ζητήματα ε, της ανθρωπιστικής ατζέντα. Πρώτον, το Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Ε, συμφωνώ με την Επίτροπο Γεώργιεβα ότι η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω του Ευρωπαϊκού Σώματος Εθελοντών εκφράζει πέρα από την παροχή της βοήθειας καθ' αυτής, την, μία από τις σημαντικότερες αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την αλληλεγγύη. Η αλληλεγγύη είναι μία από τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά επίσης και ε, θεμελιώδες στοιχείο των προτεραιοτήτων της, της Κυπριακής Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρούμε ότι αυτές τις δύσκολες εποχές όπου οι συγκρούσεις και τα προβλήματα εντείνονται. Η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Σώματος Εθελοντών για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας θα δημιουργήσει την κατάλληλη πλατφόρμα μέσω της οποίας οι νέοι της Ευρώπης θα μπορούν να εκφράσουν τη λελεγγύη τους με ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο. Όπως γνωρίζετε, οι εργασίες για την σύσταση του Ευρωπαϊκού Σώματος Εθελοντών Παροχής Ανθρωπιστικής Βοήθειας προχωρούν επιτυχώς. Ε, γνωρίζουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εκφράσει το έντονο ενδιαφέρον του για αυτό ε, το, το, εγχείρημα και έχει αποφασιστικό ρόλο να διαδραματίσει στην υλοποίησή του. Η Κυπριακή Προεδρία βασίζεται στην συνεισφορά σας έτσι ώστε να δημιουργηθεί, να ε, ιδρυθεί αυτό το σώμα αρχές φθινοπόρου. Δεύτερον, η Σύμβαση για την Επιστημιστική Βοήθεια. Όπω έχει αναφέρει και η Επίτροπο Γεώργιβα, η η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν πρωταγωνίστησε στην ανανέωση της Σύμβασης για την Επιστημιστική Βοήθεια το 1999. Ο βασικός στόχος της επαναδιαπραγμάτευση ήταν να αξιοποιηθούν πιο σύγχρονα εργαλεία επιστημιστικής βοήθειας. Ε, μια νέα σύμβαση θα μπορέσουμε να απευθυνθούμε στους πλέον ευάλωτες ε, ε, πλέον ευάλωτους ανθρώπους με τρόπο πιο αποτελεσματικό. Ο κοινό μας στόχος των θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών είναι η σύμβαση αυτή να επικυρωθεί όσο το δυνατόν πιο νωρίς, κάτι που θα δώσει ένα ισχυρό σήμα και στην διεθνή κοινότητα και στους εταίρους μας ε, όσον αφορά τη δέσμευσή μας για την παροχή επιστημιστικής βοήθειας και την επιστημιστική ασφάλεια. Θα συνεργαστούμε στενά μαζί σας προς ε, την υλοποίηση αυτού του κοινού στόχου. Τρίτον, η υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Συνένεσης για την ανθρωπιστική βοήθεια και το πρόγραμμα δράσης. Η ενδιάμεση αναθεώρηση της ε, ε, συνένεση για την ανθρωπιστική βοήθεια και του προγράμματο δράση είναι μια διαδικασία την οποία παρακολουθούμε από στενά. Στο πλαίσιο αυτό η ε, πρωτοβουλία, η γνωμοδότηση ιδίας πρωτοβουλίας που ε, συνέταξε η κυρία Στριφλέρ, μέλος της Επιτροπής σας, και υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Ιανουάριο του 2011 ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη. Η Δανική Προεδρία συνέχισε τη συζήτηση για την υλοποίηση τους ενδιάμεση αναθεώρηση και του προγράμματος δράσης ε, που αποτέλεσε την βάση για τα συμπεράσματα του ε, Συμβουλίου του Μαΐου της προηγούμενης χρονιάς μια συζήτηση η οποία έγινε στο πλαίσιο της Ομάδας Ανθρωπιστική και Επιστημιστική Βοήθεια του Συμβουλίου. Θα συνεχίσουμε λοιπόν, εκ μέρους τη Κυπριακή Προεδρία, την πολύ καλή ε, εργασία που ξεκίνησαν η Πολωνική και η Δανική Προεδρία, η Στο τέταρτο σημείο, η Ευρώπη προσπαθεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του λοιμού και του υποσυντισμού. Όπως έχει αναφέρει και η Επίτροπος Γεώργεβα, Η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας μπορεί να απαλύνει τον πόνο, αλλά δεν είναι ο τρόπος να θεραπεύσουμε την ίδια την ασθένεια. Προκειμένου να αντιμετωπίσουμε και να προλάβουμε τον υποσυτισμό και τον λοιμό στο μέλλον, θα πρέπει να συνοδεύσουμε αυτή την βοήθεια ε, με ε, βοήθεια η οποία θα βοηθά τα κράτη να αντιμετωπίσουν ε, την ξηρασία στο μέλλον. Δεν μπορεί μια προσέγγιση ad hoc ε, σε κάθε περίπτωση να είναι ε, αποτελεσματική. Έτσι λοιπόν, η ενίσχυση της ε, αντοχής ενός κράτους συνδυάζοντας την βοήθεια και την ανάπτυξη ε, προκειμένου να αντιμετωπιστούν και οι φυσικές αλλά και οι ανθρωπογενείς καταστροφές. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να προχωρήσουμε. Η καλύτερη παροχή βοήθειας μπορεί να συνεισφέρει στην ανάπτυξη και η καλύτερη ε, ε, ανάπτυξη μπορεί να βοηθήσει στην μετάβαση από τη μία κατάσταση στην άλλη. Η σύνδεση λοιπόν της ε, βοήθειας, της αρρωγής και της ανάπτυξης εκφράζεται μέσω των προετυποβλιών των επιτρόπων της Επιτρόπου Κερκίεβα και του Επιτρόπου Πίγκυπαλς Συνεχίζοντα λοιπόν αυτό την προσπάθεια και η Κυπριακή ε, Προεδρία θα προσπαθήσει να δημιουργήσει τέτοιες συνδέσεις ε, της ανθρωπιστικής βοήθειας και της βοήθειας αναπτυξιακής συνεργασίας σε χώρες που υφίστανται κρίση ή μετά από κρίση. Τώρα θα ήθελα να εστιάσω σε δύο συγκεκριμένες ανθρωπιστικές κρίσεις στη Σαχέλ και στο κέρας της Αφρικής. Αυτές οι ανθρωπιστικές κρίσεις δείχνουν πόσο απαραίτητο είναι να αντιμετωπίζουμε τους ε, λόγους που βρίσκονται πίσω, τους δομικούς λόγους που βρίσκονται πίσω από την επιστημιστική ανασφάλεια και να ενισχύσουμε τις χώρες της περιοχής. Όπως γνωρίζουμε, οι παράγοντες που δημιουργούν την το, το πρόβλημα επιστημισμού είναι οι κακές οδιές που δημιουργήθηκαν εξαιτία κλιματικών προβλημάτων. Θα ήθελα λοιπόν να συγχαρώ τους επιτρόπους Γεωργίευα και Πίγκμπαλξ για το γεγονό ότι διοργάνησαν μια συνάντηση υψηλού επίπεδου εδώ στι Βρυξέλλε σε σχέση με το Σαχέλ και την επιστημιστική κρίση. Λίγες εβδομάδες πριν φτάσουμε στο πιο δύσκολο σημείο αυτής της κρίσης, όπου προβλέπεται ότι 18 εκατομμύρια άνθρωποι θα κινδυνεύσουν από λοιμό. Είναι ε, ενθαρρυντικό να βλέπουμε πόσο ε, ευρεία εκπροσώπηση υπήρξε από τις χώρες του Σαχέλ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και την διεθνή κοινότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο ηγέτης παγκοσμίων στην παροχή ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας παγκοσμίω και είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αύξησε την ανθρωπιστική ε, βοήθεια προς το Σαχέλ κατά 40 εκατομμύρια ευρώ με αποτέλεσμα η συνολική βοήθεια προς το Σεχέλ να ε, ανέλθει στα 337 εκατομμύρια ευρώ. Όπως έχουν αναφέρει και η Επιτροπή Γεωργίευα και Πίμπαλξ, είναι πολύ σημαντικό να εστιάσουμε τους ε, παράγοντες που οδηγούν στην ε, χρόνια επισητιστική ανασφάλεια στην περιοχή του Σαχέλ. Έτσι ώστε να βοηθήσουμε αυτές τις χώρες να είναι καλύτερα προετοιμασμένες να αντιμετωπίζουν τέτοιες κρίσεις και όχι απλώς να ανταποκριθούν αποκρινόμαστε μετά την εκδήλωσή τους. Γι' αυτό είναι σημαντική η υλοποίηση της πρωτοβουλίας Αγίρ που ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σύνδεση της αρρωγής, της αποκατάστασης και της ανάπτυξης είναι μία από τις θεμελιώδεις προτεραιότητες του, στην ανθρωπιστικό τομέα της Κυπριακής Προεδρίας. Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να προχωρήσουν αυτά τα θέματα και δεν, η δέσμευσή μας δεν αφορά μόνο ε, στην παροχή βοήθειας στους ανθρώπους του Σαχέλ στην διάρκεια της τρέχουσας κρίσης, αλλά επίσης στο να τους βοηθήσουμε να σπάσουν αυτόν τον φαύλο κύκλο ε, χρόνιας επιστημιστικής κρίσης. Και για να γίνει αυτό πρέπει να αξιοποιήσουμε τη συνέργεια μεταξύ της ανταπόκρισης σε κρίση, της ε, τη ανθρωπιστικής βοήθειας και της αναπτυξιακής βοήθειας. Τώρα, όσον αφορά την πρωτοβουλία SHARE για το κέρα της Αφρική. Όλοι γνωρίζουμε τα ε, σοβαρά ανθρωπιστικά και αναπτυξιακά αλλά και προβλήματα ασφαλείας που ε, αντιμετωπίζουν οι χώρες του κέρατος της Αφρική. Πρέπει να συνεχίσουμε να τις προσπάθειες μας για να σπάσει αυτός ο φαύλος κύκλος των κρίσεων και να βοηθήσουμε τις χώρες αυτές να μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα σε καταστροφές στο μέλλον. Πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ε, κατανείμει 250 εκατομμύρια ευρώ με στόχο να βοηθήσει την προετοιμασία ανταπόκριση σε κρίσεις και την επιστημιστική ασφάλεια στις χώρες του κέρατος της Αφρικής. Η πρωτοβουλία SHARE ε, έχει στόχο να βοηθήσει τις τοπικές κοινωνίες, κοινότητες στην περιοχή να αντιμετωπίσουν την ξηρασία και άλλες φυσικές καταστροφές, βοηθώντας ε, σε τομείς όπως η διαχείριση των υδάτων, ε, η υγιεινή και ο επιστημισμός. Βλέπουμε ήδη από τα αποτελέσματα επιτόπου της πρωτοβουλίας ΣΕΡ θα συνεχίσει η Κυπριακή Προεδρία ε, τέτοιου είδους πρωτοβουλίες προκειμένου να ενισχύσουμε την ικανότητα ανταπόκρισης ε, και πρόληψης ε, τέτοιων κρίσεων σε περιοχές που κινδυνεύουν με ξηρασία. Η Κυπριακή Προεδρία επίσης το τέλος Νοεμβρίου θα διοργανώσει ένα διεθνές συμπόσιο για την ανθρωπιστική βοήθεια. Προσπαθούμε να φέρουμε στο ίδιο τραπέζι την κοινωνία των πολιτών αλλά και τους υπεύθυνου για τη χάραξη πολιτικής έτσι ώστε να ανταποκριθούμε ε, στα ζητήματα ε, της επιστημιστικής ασφάλειας. Και κλείνοντας την παρουσίασή μου για το ε, πρόγραμμα της Κυπριακής Προεδρίας για όλα τα ανθρωπιστικά ζητήματα, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω, να διαβεβαιώσω όλα τα μέλη αυτής της Επιτροπής, ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι περνάει το χέρι μας για να συνεχίσουμε την, το εξαιρετικό έργο που ήδη ξεκίνησαν οι δύο α, εταίροι μας, το τρίο της Προεδρίας, η Πολωνία και η Δανία. Θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι προσβλέπω σε μια υποκοδομητική συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συγκεκριμένα με την Επιτροπή Ανάπτυξης προκειμένου να προχωρήσουμε τις προτεραιότητες μας στην παγκόσμια ανθρωπιστική ατζέντα. Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ όλους, αγαπητά μέλη της Επιτροπής, για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε, κύρια Υπουργέ. Σας ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Ο κύριος Γκέι Μίσελ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ, και καλώς ορίσατε. Καταρχάς θα ήθελα να πω ότι χαιρόμαστε πολύ που σας βλέπουμε εδώ. Τόσο νωρίς στην Προεδρία σας και πραγματικά το εκτιμούμε τα μάλα. Δεν ξέρω αν θα μπορούσατε απαντώντας σε κάτι που θα πω σύντομα να μας πείτε δύο λόγια παραπάνω. Ε, για το Νοέμβριο δεν κατάλαβα ακριβώς τι θα διεξαχθεί εκεί. Μπορείτε να το αναπτύξετε λίγο περισσότερο για τη διάσκεψη αυτή του Νοεμβρίου. Προσπαθήσαμε να ορίσουμε προτεραιότητες κατά τη ε, ε, διάρκεια της θητείας μας, για το υπόλοιπο της θητείας και την επόμενη. Υπάρχουν ε, κάποιες προτεραιότητες που πρέπει να οριστούν, αλλά το πρόβλημα ποιο είναι. Όταν κανείς έχει πάρα πολλές προτεραιότητες, είναι σαν να μην έχει καθόλου. Και θα πρέπει να ορίσουμε κάποιες σούπερ προτεραιότητες από αυτές, αντί να προχωρούμε συνεχώς. ήθελα ενδεχομένως να σας προτείνω πρώτη προτεραιότητα να είναι η συνοχή της πολιτικής και η συνεκτικότητα, ε, καλύτερο συντονισμός δηλαδή να υπάρχει μεταξύ των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προστασία από τους κινδύνους και από τις ε, θεομηνίες και τις καταστροφές. Μιλήσατε για την ΑΕΤ. Δεν έχω τα στοιχεία μου, αλλά είναι εύκολο να το πάρουμε από τον ΟΗΕ. Εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων έχασαν τη ζωή τους από αιτήσει ομιλίες ε, θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν. Το θέμα δεν είναι να ερχόμαστε να ε, μαζεύουμε τα σπασμένα. Και σήμερα στην ΑΕΤ και αλλού ο κόσμος δεν ζει σε ασφάλεια. Και όταν έρχεται η θεομηνία, καταστρέφει τα σπίτια τους, χάνουν τις ζωές τους. Ε, θα παρακαλούσα να υπάρχει ε, μια μεγαλύτερη συνέχεια στην πολιτική μας και συνεκτικότητα για την πρόληψη των κινδύνων. Και καλό θα ήταν ενδεχομένω ως προτεραιότητα να το θέσετε υπόψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων κρατομελών για να μπορέσουν να το υιοθετήσουν και οι υπόλοιποι. Και θα πρέπει να υποσυ ε, υποστηριχθεί αυτό και από μη κυβερνητικέ οργανώσει, μικρομεσαίε ε, οργανώσεις που ασχολούνται με τα δικαιώματα των παιδιών. Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας νομίζω ότι μπορείτε εσείς να το προωθήσετε αυτό το θέμα και να γίνουν και πρόοδοι. Λοιπόν, θα σας παρακαλούσα, θα σας ρωτούσα Υπουργέ, να μας πείτε τι ακριβώς θα γίνει ε, το Νοέμβριο στην Κύπρο και θα υπάρχει δυνατότητα να προωθηθούν τέτοια θέματα στην ημερήσια διάταξη και να αποκρισταλώσουμε κάποιες σούπερ προτεραιότητες αυτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριος Γκέρετς έχει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Ο Γκέι Μίσελ νομίζω ότι ουσιαστικά θέματα ρώτησε δύο παρατήρησεις. Να ευχαριστήσω την ε, Υπουργό ε, της Κύπρου που ήρθε εδώ, απίθυνε το λόγο στην Επιτροπή μας, η πρώτη φορά που ανταποκρίνεται σε αυτή την πρόκληση η Κύπρος, ε, αξίζεται την υποστήριξή μας και της Επιτροπής μας επίσης ε, και με το ταλέντο σας επίσης, με το οποίο αναπτύξατε όλα αυτά τα προβλήματα και ε, πέρα από την ανθρωπιστική βοήθεια, την κατεπίγουσα βοήθεια, θα μπορούσατε να πείτε και περισσότερα πράγματα και για τις προτεραιότητες της ανάπτυξης, ε, αν θέλετε εδώ να πείτε αυτά τα πράγματα, πάντως θα σας ακούγαμε ιδιαίτερα προσεκτικά. Κύριε Μπέρμαν, έχετε το λόγο. Thank Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι οι Επίτροποι Γεωργίευα και Πίπαλξ διοργάνωσαν αυτή τη διάσκεψη Βρυξέλλες για το Σαχέλ, όπου υποσχέθηκε ότι θα έχουμε κοινή προσέγγιση για όλα αυτά τα προβλήματα που έχει η περιοχή και ανασφάλειας και από κοινού να προλαμβάνουμε τέτοιες καταστάσεις να επαναληφθούν όλοι μαζί οι δωρητές, ε, η UNICEF, ε, η UNDP και οι χώρες ήδη στη Σαχέλ και άλλοι. Ε, ωστόσο, ακόμα και αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει 340 εκατομμύρια ευρώ φέτος στο Σαχέλ, ο αριθμός των παιδιών που αναμένεται να πεθάνουν από υποσυντισμό φέτος και μόνο είναι 300.000. Και τα μισά στο τσάτ και μόνο. όλη αυτή η αποφασιστική δράση δεν αποτρέπει τις ομιλίες από το να συμβαίνουν, αλλά θα πρέπει ε, πραγματικά να ευχαριστήσουμε και να ποτίσουμε φόρο τιμή στους επιτρόπους για αυτή την αποφασιστική τους στάση. Θα ήθελα ε, να σας ευχαριστήσω που ήρθατε τόσο νωρίς ε, από την ανάληψη της Προεδρίας στην Επιτροπή μας, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα ανάμεσα στις πολιτικές της ανάπτυξης και την ανθρωπιστική δράση ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο πρόβλημα στην εκταμείευση των πόρων. Ε, κλασικά η ανθρωπιστική βοήθεια δίνεται πάρα πολύ γρήγορα, διότι λειτουργούν σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και είναι και συνηθισμένοι οι άνθρωποι αυτοί στις διαδικασίες ταχύτατης εκταμείευσης, ενώ η αναπτυξιακή πολιτική κατεξοχήν χρειάζεται περισσότερο χρόνο. Αυτά τα δύο δεν ταιριάζουν. Ε, και επιτόπου είναι πρόβλημα γιατί δεν μπορούν να συντονιστούν. Και το έχω ρωτήσει επανειλημμένα σε πολλούς και από ό,τι φαίνεται το πρόβλημα ακόμα δεν έχει λυθεί. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, αν συνδέσετε αυτά τα τρία, τη βοήθεια, την αποκατάσταση και την ανάπτυξη, ε, ως προτεραιότητα της Προεδρίας σας μπορείτε να φροντίσετε οι διαδικασίες εκταμίευσης ακριβώς σε αυτές τις δράσεις που στόχο έχουν την ενίσχυση ε, τις σχέσεις αρρωγής με ανάπτυξη, να είναι τέτοιες οι διαδικασίε εκταμίευσης, ώστε να υπάρχει αυτό ο σύνδεσμο και να είναι πραγματικότητα. Και ένα δεύτερο που θα ήθελα να σα ρωτήσω είναι το θέμα ε, της ανθεκτικότητας ε, του πληθυσμού σε περιοχές που υφίστανται καταστροφές και θεομηνίες. Αυτό έχει να κάνει πολύ με κάποιες πολιτικές που αρχίζουν από το σεβασμό του ντόπιου πληθυσμού. Αν στην Αιθιοπία, Φερρυπίν, η κεντρική κυβέρνηση δεν σέβεται ε, ε, εκείνους που ζουν στο Νότο, ε, ποτέ δεν πρόκειται να υπάρχει ανθεκτικότητα για αυτούς τους πληθυσμούς και πρόληψη. Παίζουν όμως πολύ σημαντικό ρόλο για την παραγωγή τροφίμων στο Σαχέλ αυτοί οι βοσκοί που ζουν στην Νότια Αιθιοπία, γιατί ε, έχουν και τα κοπάδια τους εκεί και, είναι μια τοπική κοινωνία. Χρειάζεται λοιπόν πολιτική δράση, όχι μόνο στην Αιθιοπία και στην πρωτεύουσα, αλλά και στον Αϊρόμπι. Έτσι ώστε οι ντόπιοι πληθυσμοί να βλέπουν τα δικαιώματά τους να γίνονται σεβαστά και να συνεχίσουν να ζουν με τον τρόπο που παραδοσιακά θέλουν, ε, με τον πολιτισμό τους κτλ. Αυτό όμως αντιτίθεται ε, σε κάποιες αλαζονικές ιδέες του αστικού πληθυσμού ότι αυτοί οι βοσκοί εκεί πέρα ζουν ε, με υπομεσαιωνικές συνθήκες και θα πρέπει πολύ γρήγορα να εξυγχρονιστούν, να γίνουν τεχνοκράτες και να ευθυγραμμιστούν με την πόλη. Αυτό δεν ισχύει. Μπορεί να υπάρχει κάποιο μέση οδός. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει και η Πρόεδρος. Και τώρα μου παραχωρώ το λόγο. Σημείωσα το ενδιαφέρον σας για την ανθρωπιστική βοήθεια, όπως επίσης και τις προτεραιότητες που αποδίδεται. Αλλά παρακαλώ προσέξτε ότι στο σχέδιο προϋπολογισμού 2013 και για τα επόμενα χρόνια ο προϋπολογισμός είναι μειωμένος ε, για την ανθρωπιστική βοήθεια και κυρίως τα κονδύλια για την Παλαιστίνη μειώθηκαν ιδιαίτερα ενώ υπάρχουν ακόμα περισσότερες ανάγκες. Αυτή είναι η πρόταση του Συμβουλίου και το Κοινοβούλιο. Στο Κοινοβούλιο προσπαθούμε να διορθώσουμε κάπως τα πράγματα και εμεί στην Επιτροπή Ανάπτυξης προτείνουμε μια αύξηση αλλά θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας ότι έχει προτεραιότητα αυτή η πολιτική και ότι υπάρχουν πολλά και διάφορα τα οποία όμως δεν μας επιτρέπουν ακριβώς να μειώσουμε τα κονδύλια που πάνε εκεί. Η κυρία Θεοχάρους έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα με τη σειρά μου να καλωσορίσω την έντιμη Υπουργό Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας την ε, οποία γνωρίζω από τα φοιτητικά μας χρόνια όταν μαζί κάναμε αγώνες για την δημοκρατία μαζί κάναμε αγώνες για την δημοκρατία στην Ελλάδα σε μια περίοδο που ήταν πάρα πολύ δύσκολο να τολμά κανείς να πει την άποψή του. Η κυρία Υπουργός ήταν πολύ σεμνή και πολύ ντροπαλή θα έλεγα στην παρουσίαση των θεμάτων, αλλά έχει μια σημαντική δράση στην χώρα μας που πραγματικά θα άξιζε τον κόπο να τη γνωρίζουν οι συνάδελφοι. Πρέπει να σας πω ότι η Κύπρος είναι η μόνη χώρα από τις νέες που καλύπτει το 0,7 του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος σε αναπτυξιακή βοήθεια. Η Κύπρος παρά τα προβλήματα τα οποία έχει όντας μια χώρα υποκατοχή και μάλιστα σκληρή κατοχή με το 1 τρίτο του εδάφους της κατεχόμενο και με το 1 τρίτο του πληθυσμού της ε, να ζει σε προσφυγικούς οικισμούς έχει καταφέρει να είναι μια πραγματική ε, ανθρωπιστική υπερδύναμη έχοντας, ανθρωπιστική, έχοντας στείλει ανθρωπιστική βοήθεια σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου που συνίστανται σε επισητιστική βοήθεια, σε αναπτυξιακή βοήθεια, σε ε, δεντροφιδεύσεις, αναδασώσεις, στην προσπάθεια της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, της απερίμωσης, στέλνοντας ειδικού γεωλόγους και ε, γεωπόνους σε όλες τις υποανάπτυκτες χώρες, δίνοντας υποτροφίες και εκπαιδεύοντας νέα παιδιά να γίνουν μαμές, να γίνουν νοσοκόμες, να εκπαιδευτούν στην ιατρική, στο, στα δασικά μας κολέγια, στα γεωργικά κολέγια. Η Κύπρος έχει μία παράδοση σε αυτό το θέμα. Θα μπορούσε να γίνει το κέντρο της περιφερειακής βοήθειας ή στην Ανατολική Ευρώπη. Να σας θυμίσω με ποιο τρόπο η Κύπρος χειρίστηκε θαυμάσια την ανθρωπιστική κρίση του Λιβάνου όταν έπρεπε να γίνει ε, εκένωση του Νότιου Λιβάνου από τον πόλεμο ε, το 2006. Συμφωνώ με την κυρία Πρόεδρο ότι στο επόμενο, στην επόμενη περίοδο 2014-2020 θα υπάρχουν μικρότερα ε, ε, κονδύλια για να διατεθούν. Όμως, κυρία Πρόεδρε, έχει τεράστια σημασία η σωστότερη διαχείριση αυτών των κονδυλίων. Με σωστότερη διαχείριση θα έχουμε τα ίδια αποτελέσματα αν αποφευθούν οι, δαπάνε, οι σπατάλες και αν αποφευθεί η διαφθορά εκείνη που προέρχεται από διεφθαρμένα καθεστώτα κυβερνήσεις και ε, τοπικές κυβερνήσεις. Άρα ο συντονισμός είναι εκείνος ο παράγοντας ο οποίος θα δημιουργήσει και την ειδοποιώ διαφορά και οι κυβερνήσεις μαζί με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και την κοινωνία των πολιτών σίγουρα θα φέρουν καλύτερο αποτέλεσμα γιατί εμείς στηριζόμαστε στην κοινωνία των πολιτών. Έχω δύο ερωτήσεις προς την κυρία Υπουργό. Η μία είναι αν προτιθέμεθα να στηρίξουμε την προσπάθεια δημιουργίας ανθρωπιστικής δύναμης άμεσης παρέμβασης Humanitarian Task Force που είναι εντελώς διαφορετικό από το συντονιστικό όργανο των εθελοντών στο οποίο προσανατολίζεται η κυρία ε, Εκείνο που χρειάζεται είναι να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης και καταπελτικής αντίδρασης μέσα στο πρώτο 24ωρο κατά το οποίο θα εκδηλωθεί μια καταστροφή και θα μπορούσε να γίνει αυτό με δύο ή τρία κέντρα σε όλη την Ευρώπη. Δεν είναι απαραίτητο να ξεκινά από την Ευρώπη να πηγαίνουν στην άλλη μεριά του κόσμου, στην ΑΕΤ, αλλά άνετα η Ευρώπη θα μπορούσε να καλύψει το πρώτο 24ωρο την Αφρική, δηλαδή να βλέπουμε και τα μεγέθη. Το ίδιο ισχύει βέβαια όσον αφορά τα ζητήματα των μεγεθών και για τι δυνατότητε που έχει η κάθε χώρα να προσφέρει. Και δεύτερον, κυρία ε, Υπουργέ, θα ήθελα να σα ρωτήσω αν αληθεύει ότι έχετε προτείνει την κυβέρνησή σας ένα τμήμα από τα ενδεχόμενα κέρδη που θα έχει Κύπρος από την εξόριξη του φυσικού αερίου να διατίθεται αποκλειστικά για αναπτυξιακή βοήθεια προς όφελος των τρίτων χωρών. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Στίφλερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ. Συγγνώμη, συγγνώμη που καθυστέρησα, αλλά ψηφίζαμε για... με καθυστέρηση πάνω από ώρα και δεν μπόρεσα να έρθω νωρίτερα. Δεν πίζω να μου πούν τι έγινε εδώ μεταξύ κατά τη διάρκεια της απουσίας μου, αλλά για αυτό το εθελοντικό σώμα μια ερώτηση. Υπάρχουν διάφορες αμφιβολίες, αντιδράσεις από το Συμβούλιο. Εσείς ε, πώς θέλετε να διαχειριστείτε το όλο θέμα η άποψή σας σχετικά ποια είναι. Και όπως είπε πριν από λίγο η κυρία Θεοχάρους, θα ήθελα να αναγνωρίσω τη συμβολή της Κύπρου και ελπίζω ότι η Προεδρία σας θα μας βοηθήσει να δώσουμε το παράδειγμα και σε άλλες χώρες που δυσκολεύονται και θα μπορούσαν να συνεισφέρουν περισσότερο. Αυτό κυρίως σχετικά με αυτό το εθελοντικό σώμα πολιτικής προστασίας. Ο έχει ε, Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας και εγώ είμαι πεπισμένος ότι η Κύπρος ε, θα διαδραματίσει θετικό ρόλο στην ανθρωπιστική βοήθεια. Έχετε το πλεονέκτημα να βρίσκεστε πολύ κοντά ε, στις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και έχετε και την ανάλογη ευαισθησία γιατί εδώ και γενναίες αυτές οι συγκρούσεις έχουν τον αντίκτυπό τους και στην ε, Κύπρο. Αναφερθήκατε στην Παλαιστίνη και την ανθρωπιστική βοήθεια, ιδιαίτερα στη λωρίδα της Γάζας, που είναι αμέσως απέναντι από την Κύπρο. Η ανθρωπιστική κατάσταση από χρόνο σε χρόνο επιδεινώνεται. Είναι μια περιφέρεια που πριν από λίγα χρόνια μπορούσε να έχει αυτάρκεια στα τρόφιμα και τώρα ε, κατά τα μισά τρόφιμα εξαρτάται από το Ηνωμένα Έθνη για την παροχή επιστηστικής βοήθειας. Και προσβλέπω πολύ στην Προεδρία σας και ε, με την τετραμερή για την ε, Μέση Ανατολή και την κυρία Άστον να δραστηριοποιηθείτε για να βελτιωθεί η ανθρωπιστική κατάσταση ιδιαίτερα στη Λωρίδα της Γάζας. Ευχαριστώ. Τώρα η κυρία Παπαδοπούλου παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ με τη σειρά μου να καλωσορίσω την κυρία Μαρκουλή, την Υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου. Να πω ότι ε, σήμερα είχαμε μια δύσκολη μέρα γιατί είχαμε πολλές ψηφοφορίες. Γι' αυτό και εγώ δεν μπόρεσα να παρακολουθήσω από την αρχή την παρουσίασή της. Οι ερωτήσεις με επικεντρώνονται σε δύο ερωτήματα. Πριν από λίγο συζητούσαμε στην Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων μια γνωμοδότηση που αφορούσε ακριβώ την κύρια επιτροπή, την Επιτροπή Ανάπτυξη. Και είχαμε εντοπίσει ότι υπάρχουν πολύ ψηλά ποσοστά μητρική και παιδική χρησιμότητα που είναι δυσανάλογα ψηλά στι αναπτυσσόμενε χώρε. Και ακριβώ ανάμεσα στα πολλά ανθρωπιστικά προβλήματα που συναντούν οι γυναίκε σε αυτέ τι χώρε και τα παιδιά, προκύπτει ιδιαίτερα μεγάλη ανάγκη για να παρέχεται υψηλή προστασία επίγουσα με ευτική περίθαλψη, όπως επίσης να μειωθούν τα ποσοστά της μητρικής και της παιδικής θνησιμότητας. Κοντά σε αυτά είχαμε μιλήσει για το γεγονός ότι πολλές γυναίκες στις αναπτυσσόμενες χώρες στερούνται βασικής ενημέρωσης όσον αφορά σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία. Και επίσης ε, είναι θύματα γιατί παραβιάζονται πολλά ανθρώπινα δικαιώματα είναι θύματα εξαναγκασμών σε γάμους σε πολύ νεαρή ηλικία, ακροτηριασμού των γεννητικών οργάνων ε, και όλα αυτά οπωσδήποτε είναι και απότοκο της εκτεταμένης βίας που είναι πολλές φορές απότοκων έφυλων ανισοτήτων. Και η εισήγηση που θα κάνει η Επιτροπή Γυναικών προς την Επιτροπή Ανάπτυξης είναι ακριβώς να τεθεί ως προτεραιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της πολιτικής της για την αναπτυξιακή βοήθεια η καταπολέμηση της ατιμορρησίας των δραστών των ελόγων βιοπραγιών που γίνονται εναντίον των γυναικών στις αναπτυσσόμενες χώρες και να γίνουν ακριβώς περισσότερα προγράμματα ενημέρωσης ώστε οι γυναίκες να ξέρουν τα δικαιώματά τους και να τα διεκδικούν. Θα ήθελα να μου πείτε αν στη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας θα μπορούσε να ακριβώς να πιέσει η Κυπριακή Προεδρία προς αυτήν την κατεύθυνση. Να γίνει δηλαδή προτεραιότητα ε, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής πολιτικής για βοήθεια η καταπολέμηση της ατιμορρησίας των δραστών για βιοπραγίες εναντίον γυναικών. Και η δεύτερη ερώτηση αφορά ακριβώς το γεωστρατηγικό ρόλο της Κύπρου. Η Κύπρος είναι το νοτιότερο σημείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που γειτονιάζει με τις χώρες της Μέσης Ανατολής. Έχει πράγματι μια παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας και πολλές φορές ακούοντας κάποιους συναδέλφους να βλέπουν με υποτιμητικών τρόπο την ανάληψη της, της Κυπριακής Προεδρίας από μια μικρή χώρα η οποία βιώνει την κατοχή, ε, ένιωσα την ανάγκη να υπερασπιστώ τη χώρα μου γιατί έχει αποδείξει όλα τα χρόνια ότι μπορεί να προσφέρει πολλά στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας. Διερωτούμε, θα μπορούσε ε, να γίνει ένας οργανισμός ευρωπαϊκός στην Κύπρο, ο οποίος ακριβώς λόγω της γυτνίασης με αυτές τις χώρες που έχουν προβλήματα, να είναι ο ευρωπαϊκός εκείνος οργανισμός που να στηρίζει κάθε βοήθεια και ανθρωπιστική και άλλη μορφή, και ουσιαστικά να εδρεύουν εκεί άνθρωποι εμπειρογνώμονε που να στηρίζουν τις γειτονικέ μας χώρες σε περιπτώσει και φυσικών αλλά και άλλων καταστροφών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Υπουργό τώρα έχει το λόγο για να μπορέσει να μας απαντήσει στα ερωτήματα που έθεσαν τα μέλη της Επιτροπής Ανάπτυξης. Merci, Madame la ε, First of all, uh, let me... Uh, Σας ευχαριστώ πολύ. Επιτρέψτε μου να πω μερικά λόγια ακόμα για το Διεθνές Συμπόσιο που θα διεξαχθεί στην Ευκοσία ε, 23 ε, Νοεμβρίου με τίτλο «Ένα πλαίσιο με κινητήρια δύναμη τους ε, πολίτες μετά το 2015». Το διοργανώνει μια πλατφόρμα πανκύπρια μη κυβερνητικών οργανώσεων. Και πρέπει να σας πω ότι είναι μια πρωτοβουλία ε, από πλατφόρμες ελληνοκυπριακές και τουρκοκυπριακές ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις που διοργανώνουν αυτό το συμπόσιο με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στα πλαίσια της παγκόσμιας πρωτοβουλίας προς ένα νέο πλαίσιο αναπτυξιακό μετά τους στόχους της χιλιετίας μετά το 2015 αποφασίσαμε να συμπεριλάβουμε και τη συζήτηση για το πρόγραμμα μετά τους αναπτυξιακούς στόχους της ε, χιλιετίας και είναι βασικό στοιχείο της ε, Προεδρίας μας. Η Κύπρος θα συνδεθεί με τη Διεθνή Εκτελεστική Επιτροπή και θα υποδεχτεί διεθνές συμπόσιο με θέμα τη συζήτηση μετά το 2015, το Δεκέμβριο του 2012, με στόχο να ολοκληρωθούν οι εθνικές διαβουλεύσεις και να έχουμε μια συνολική θέση της κοινωνίας των πολιτών για τη συζήτηση μετά ε, τους στόχους της χιλιετίας. Εκεί θα συμμετέχουν εκπρόσωποι από την Ευρώπη αλλά και παγκοσμίω και από την κοινωνία των πολιτών, καθώ επίσης και εκείνοι που παίρνουν τις αποφάσεις. Ε, η Κύπρος δεν θα διοργανώσει τις Ευρωπαϊκές ημερίδες ε, ανάπτυξης. Αυτό το συγκεκριμένο γεγονός φιλοδοξεί να καλύψει το κενό που ε, δημιουργείται από αυτό το υψηλό επίπεδο και πολύ προβεβλημένο γεγονός τους. Ε, σε αυτή τη διημερίδα θα ακούσουμε ιστορίες, εκθέσεις ε, και θα δούμε πώς θα μπορέσουμε να διαμορφώσουμε ένα αποτελεσματικό πλαίσιο για την εξάλληψη της φτώχειας. Για να συνδεθεί αυτό με τις Ευρωπαϊκές ημερίδες περιβάλλοντος Βρυξέλλης και με τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας, ε, μία από τις βασικές θεματικές ενότητες του Συμποσίου θα είναι η επιζητιστική ασφάλεια ε, ε, διαδραστικές συνεδριάσεις των ομάδων εργασίας θα μας επιτρέψουν να διερευνήσουμε διάφορα ενδεχόμενα και τελικά θα προβούμε σε συστάσεις για τη διεθνή κοινότητα. Σε ό,τι αφορά την συνοχή ε, και συνεκτικότητα των πολιτικών, κύριε Μίτσελ, των αναπτυξιακών, συμφωνώ απολύτω ότι είναι άκρο σημαντικό αυτό. Η συνεργασία μεταξύ κρατών μελών δηλαδή, αλλά και το να θέτουμε αυτά τα ζητήματα υπόψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πολύ σημαντικό. Σε πρώτη ευκαιρία θα τα θέσω υπόψη ε, του Επιτρόπου κυρίου Πίμπαλξ, Είχα ήδη ε, κάποιες προκαταρτικές συζητήσεις ε, όταν ήρθε στην Κύπρο ο ίδιος. Θα το συνεχίσουμε και είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε αυτά τα θέματα νωρίτερα και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι θα δώσω συνέχεια και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Όχι μόνο να παρέχεται αυτή η ανθρωπιστική αρρωγή, αλλά να βοηθούμε και τις κοινωνίες της χώρες αυτές να οικοδομούν την απαραίτητη υποδομή για να μπορούν να προλαμβάνουν ή να ελαχιστοποιούν τις καταστροφές από τις θεομηνίες και τις συνέπειες τους. Σας ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξη, κύριε Γκέρενς για την Κυπριακή Προεδρία και νομίζω θα τη χρειαστούμε. Και χαίρομαι πάρα πολύ για την υποστήριξή σας. Σε ό,τι αφορά τη διάσκεψη για το Σαχέλ, είναι πολύ νωρίς να κάνουμε τώρα μία αποτίμηση και αξιολόγηση ε, Υποστηρίζουμε ολόθερμα την πρωτοβουλία αυτή και θα φροντίσουμε κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας τα συμφωνηθέντα στις Βρυξέλλες κατά τη διάρκεια της υψηλού επίπεδου αυτής της διάσκεψης να ε, υλοποιηθούν. Το γεγονός ότι χάνουμε ακόμα ζωές και μάλιστα πεθαίνουν τα παιδιά από υποσυτισμό και πολλές άλλες αιτίες και συνέπειες της φτώχειας και του υποσυτισμού και του λοιμού σε πολλά μέρη του κόσμου, δεν είναι ε, λόγος να μας αποθαρρύνει από το να συνεχίσουμε τέτοιες πρωτοβουλίες. Σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες εκταμίευσης, συμφωνώ απολύτως ότι θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι όταν χρειάζονται τα κονδύλια αυτά διατίθενται ε, ακριβώς εγκαίρως. Αυτά τα θέματα θα μας απασχολήσουν στο Συμβούλιο και πάλι θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι ως Προεδρία θα το συζητήσουμε με τους αρμόδιους επιτρόπους και τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να βεβαιωθούμε ότι οποιαδήποτε προβλήματα που αφορούν την εκταμείευση των πόρων που ε, είναι τόσο αναγκαίοι για τα αναπτυξιακά έργα και προγράμματα θα γίνεται γρήγορα. Σε ό,τι αφορά την ε, αντίσταση και την ανθεκτικότητα των πληθυσμών, συμφωνώ απολύτως Όταν κανείς θέτει στόχους και τους ε, προωθεί με συνέπεια σε διάφορες χώρες, σε αναπτυσσόμενες χώρες όλο τον κόσμο, πρέπει να σεβόμαστε πλήρως τον τόπιο πληθυσμό κάθε φορά, τα ήθη, τα έθιμά του και τον τρόπο με τον οποίο ε, ζει καθημερινά. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο τουλάχιστον ως Κύπρος σεβόμαστε πλήρως και θα πρέπει να πείσουμε όλους τους μεγάλους δωρητές ε, ε, προς αυτή την κατεύθυνση. Να σέβονται πλήρως τις τοπικές κοινωνίες, ε, τις κοινότητες, τα ήθη και τις παραδόσεις τους και τα έθιμά τους. Κυρία Πρόεδρε σε ό,τι αφορά τώρα τον προπολογισμό, οποιαδήποτε μείωση του προπολογισμού ανθρωπιστικής βοήθειας ε, θεωρείται απαράδεκτη, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη τις πάρα πολύ δεινές ε, συνθήκες ε, ανθρωπιστικές που επικρατούν σε πολλά μέρη, ακριβώς λόγω της κλιμάκωσης των σειράξεων ή λόγω των κλιματικών αλλαγών και των συνθήκων αν τον κόσμο. Οπωσδήποτε θα πρέπει αυτό το θέμα να μας απασχολήσει και σε καμία περίπτωση δεν θα επιτρέψουμε μείωση του προπολογισμού. Σε ό,τι αφορά το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, θα φροντίσουμε κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας στι συζητήσεις σε αυτό το συγκεκριμένο τομέα να μην υπάρξει ε, περιστολή και περικοπή στον προϋπολογισμό. Ε, ε, ε, η Ελέη είναι σπουδαία συνάλφος και μεγάλη συμπατριώτησα και θέλω να την ευχαριστήσω. Συνεχίζεται ο αγώνας μας και έχεις αποδείξει και έχουμε αποδείξει ότι η μικρή Κύπρος μπορεί να συνεισφέρει όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο, όχι μόνο στο εσωτερικό της χώρας μας, αλλά εσύ ε, η ίδια ε, στον τομέα σου έχεις επιτελέσει πάρα πολύ σπουδαίο έργο και διεθνώς και παγκοσμίως. Σε ό,τι αφορά τις προτάσεις σου για μια ανθρωπιστική ομάδα δράσης, task force, νομίζω ότι είναι σπουδαία ιδέα, θα πρέπει να κοιτάξω πώς η ιδέα αυτή και αν μπορεί να συζητηθεί περαιτέρω και μετά να λάβει τη μορφή μιας πιο ουσιαστικής πρότασης. Προσπαθήσω να συνεχίσω αυτή τη συζήτηση με εταίρους και συναδέλφους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να δούμε αν υπάρχει δυνατότητα να δώσουμε συνέχεια σε αυτή την πρόταση. Για τους υδρογονάνθρακες. Είναι πολύ νωρίς βεβαίως να κάνουμε κάποια εκτίμηση για ε, το συνολικό ποσό και ποσότητα και πόσο θα είναι το όφελος για την Κύπρο από τη νέα αυτή ανακάλυψη. Πάντως θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα ταμείο το οποίο θα καλύπτει τις ανάγκες ε, του πληθυσμού στην Κύπρο για τις επόμενες γενναίες και σίγουρα ένα τμήμα θα και μάλιστα σημαντικό θα δίνεται και στην ανθρωπιστική βοήθεια και στην απτυξιακή βοήθεια για τους λαούς και τις χώρες που το χρειάζονται. Και θα συνεισφέρουμε οπωσδήποτε στην κατεύθυνση αυτή με τρόπο ε, ουσιαστικό και σημαντικά αυξημένο και με χαρά θα το κάνουμε. Βεβαίως Χρειάζεται κάποιος χρόνος για να είμαστε σε θέση να δρέψουμε πραγματικά τους καρπούς αυτής της νέας ανακάλυψης. Αλλά είμαστε αποφασισμένοι να το πράξουμε. Για το εθελοντικό σώμα. Ε, εξ όσων γνωρίζω είναι περισσότερη υποστήριξη και λιγότερες οι επιφυλάξεις. Θα πρέπει να βρούμε τώρα έναν τρόπο να εγκρίνουμε την απαραίτητη νομοθεσία για να συσταθεί αυτό το σώμα εθελοντών και ως Προεδρία βεβαίως θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βεβαιωθούμε ότι αν υπάρχουν οποιασδήποτε επιφυλάξεις ε, και δισταγμοί των κρατών μελών να ξεπεραστούν, να αρθούν και να συνεχίσουμε την προσπάθεια αυτή και να συσταθεί αυτό το τόσο σημαντικό, εξαιρετικά σημαντικό νέο σώμα. Σε ό,τι αφορά ε, τη Μέση Ανατολή και τη Λωρίδα της Γάζας, συμφωνώ απολύτως με την ανάγκη να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή στην ανθρωπιστική κατάσταση στην Παλαιστίνη και στα κατεχόμενα εδάφη αλλά κατά κύριο λόγο στη λωρίδα της ε, Γάζας και κατά προτεραιότητα. Ε, και φυσικά ε, η Κύπρος, λόγω της μακράς σχέσεως που έχει με τις χώρες της Μέσης Ανατολής, είναι ιδιαίτερα εξαιρετικά ευαίσθητη για αυτά τα θέματα και τα τεκτενόμενα στην άμεση γειτονία μας συνεργαζόμαστε με την ύπατη εκπρόσωπο και είχα την χαρά και την τιμή να την υποδεχθώ πριν από λίγες μέρες. Είχα μακρά συζήτηση για το πώς θα μπορούσε να βοηθήσει η Κύπρος την ύπατη εκπρόσωπο και την υπηρεσία εξωτερικής δράσης σε διάφορες πρωτοβουλίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και ένας από τους τομείς ανησυχίας είναι βεβαίως το θέμα των Παλαιστινιακών εδαφών, αλλά και ο Λίβανος. Και θα προσπαθήσουμε όσο μπορούμε να βοηθήσουμε και προς την κατεύθυνση αυτή. Κυρία Παπαδοπούλου, αυτά που είπατε νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικά. Δεν είμαι βέβαιη αν αυτό το συγκεκριμένο στοιχείο έχει ληφθεί υπόψη μέχρι στιγμής στην αναπτυξιακή μας βοήθεια. Πάντως είναι εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο, αλλά και εξαιρετικά σοβαρό και ταυτόχρονα τραγικό ζήτημα. Το θέμα και η κατάσταση των γυναικών σε πολλές ε, χώρες του κόσμου, σε ό,τι αφορά την υγεία τους, αλλά και ε, τη βία κατά των γυναικών. Οπότε Οπωσδήποτε είναι και αυτό ένα θέμα το οποίο χρειάζεται ε, περισσότερη εξέταση, ε, μελέτη, αλλά κυρίως δράση για να υποστηρίξουμε τις γυναίκες αυτές και να τις βοηθήσουμε και να συνδέσουμε ως πρωτοβουλία την αναπτυξιακή βοήθεια και ε, την ανθρωπιστική βοήθεια ε, με τη θέση των γυναικών σε αυτές τις περιοχές. Δεν ξέρω αν ξέχασα τίποτα, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα πλήρες. Προτείνω, κυρία Πρόεδρε, ε, να απαντήσετε και στη Μισελ Στριφλέρ που ήρθε. Α, συγγνώμη, να επαναλάβετε τα καλά λόγια που είπατε για την κυρία Στριφλέρ στην αρχή της παρουσίασής σας, την οποία και ευχαριστήσατε. Α, ναι, ναι. Intervention. Yes. Thank you. Well. So, allow me to, to thank you. Επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω, κυρία Υπουργέ, λέει Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ και πάλι ε, που ήρθατε στην Επιτροπή μας. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε και μας υποστηρίζετε. Δείχνουμε ιδιαίτερα ευαισθησία εκεί και στο κέρας Αφρικής και στη Σαχέλ για τα θέματα αυτά, όπως επίσης για τη μάχη που δίνεται με τα προγράμματα ακριβώ κατά της πείνας ε, και σας ευχόμαστε κάθε καλή τύχη κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας. Ελπίζουμε δε ε, τους, μέσα στους επόμενους 6 μήνες της Προεδρίας σας να σας δούμε και πάλι, να σας έχουμε και πάλι ανάμεσά μας. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Α, την ημερομηνία της επόμενης συνάντησης, 3 Σεπτεμβρίου και στο ξεκίνημα έχουμε και κλεισμένο το μια, τα μέλη αμέσως μετά μια συνάντηση για λίγα λίγα λεπτά τώρα. 3 Σεπτεμβρίου 3 με 6,5 και 17 Σεπτεμβρίου από 3 μέχρι 6,5. Πέρα συνεδρίαση.